Good afternoon. Please be welcome. Καλησπέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. Και θα ήθελα να καλωσορίσουμε τους δύο υφυπουργούς από τη Σουηδία που έχουμε μαζί μας, οι οποίοι μας τιμούν σήμερα το απόγευμα με την παρουσία τους εδώ. Θα καλύψουμε μαζί του το σημείο 27 της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με την προετοιμασία από την Προεδρία του Συμβουλίου του προγράμματος της Στοκχόλμη στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα είναι αυτό το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που αποτελεί συνέχεια του προγράμματος της Χάγης στα πλαίσια της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και των ιστορικών υποθέσεων. Θα θέλαμε να ακούσουμε πρώτα τον Υφυπουργό Μάγνους Γκράνερ, που είναι αρμόδιος για ζητήματα δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων και στη συνέχεια θα ακούσουμε την κυρία Μίνα Λούγκρεν, αρμόδια για ζητήματα πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για το γεγονός ότι με προσκαλέσατε και αυτό για να συζητήσω μαζί σας προπακα... την προπαρασκευή της ε, Στοκχόλμης ε, και το πρόγραμμά μας. Αυτό το νέο πενταετές πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο θα συνεχίζει στο υφιστάμενο πρόγραμμα της Χάγης, είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της Σουηδικής Προεδρίας. Έχουμε έντονο φθινόπορο που μας περιμένει και πολλή δουλειά θα κάνουμε. Και εγώ και η συνάδελφός μου το Σεπτέμβριο μια ολόκληρη σειρά διμερών συζητήσεων και επαφών είχαμε με τα περισσότερα κράτη-μέλη ήρθαν οι εκπρόσωποι τους στη Στοκχόλμη για να συζητήσουν το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Αυτές οι διμερείς επαφές και διαβουλεύσεις ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Μας επέτρεψαν να καταλάβουμε ποιες είναι οι θέσεις των κρατών μελών και οι απόψεις τους. Η εντύπωσή μου από τις συζητήσεις σε αυτό το διμερές επίπεδο ήταν στο διμερές εκάστοτε επίπεδο ήταν ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία όσον αφορά τις ε, κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική συνεργασία και τη μελλοντική στοχοθέτηση. Έργο της Προεδρίας είναι τώρα να λάβει υπόψη αυτές τις απόψεις και να μεριμνήσει ώστε αυτές στο πρόγραμμα, στο σχέδιο προγράμματος το οποίο εμείς θα υποβάλουμε να συμπεριλαμβάνονται και έτσι να υπάρξει ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα τέλη Οκτωβρίου η Σουηδική Προεδρία θα έχει ένα πρώτο σχέδιο, πρώτο σχέδιο κειμένου που θα υποβληθεί. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εντονότερες διαβουλεύσεις μέχρι την Σύνοδο Κορυφής και την έγκριση το Δεκέμβριο. Σε αυτές τις διαδικασίες και διεργασίες φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα είναι παράγοντας που θα έχει σημασία κλειδιού για τη διαδικασία. Η Σουηδική Προεδρία είχε ήδη διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, συναντήσει, τις συνάντησε και χαιρόμαστε για την περαιτέρω καλή συνεργασία και τις, ε, την ανάπτυξη των επαφών αυτών κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Θα ακούσουμε τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα λάβουμε υπόψη τις προτεραιότητες ε, για το επόμενο πρόγραμμα για τις εργασίες τη στοκχόλμη και αναμένουμε και την πρόταση ψηφίσματο τον Νοέμβριο. Η Σουηδική κυβέρνηση επιθυμεί το πρόγραμμα της Στοκχόλμης να είναι φιλόδοξο μακροπρόθεσμο ορίζοντα να έχει χρονικά και να είναι ισορροπημένο, ισόρροπο. Πρέπει να είναι φιλόδοξο, κατά τούτο δηλαδή, καθώς εδώ σαφείς πολιτικές προτεραιότητες και πλαίσια πρέπει να τεθούν για αυτά τα οποία θέλουμε να επιτύχουμε. Τώρα, μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα πρέπει να έχει έναν φιλόδοξο χρονορίζοντα το πρόγραμμα, ώστε μακροπρόθεσμα να διαδραματίσει ένα ρόλο στην ενισχυμένη συνεργασία. Και αυτό πέρα από τα, και πάνω από τα πέντε χρόνια, πέρα και πάνω από την πενταετή περίοδο. Και ισορροπημένο επιπλέον. Ισορροπημένο, ισόρροπο, διότι στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να αποκατασταθεί μια ισορροπία, να διασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ μέτρων καταστολής η δίωξη και μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων των ε, προσώπων, των πολιτών δηλαδή και των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Αφετηρία της εργασίας αυτής, των εργασιών αυτών, ήταν φυσικά η προοπτική και η άποψη των πολιτών. Η μελλοντική συνεργασία πρέπει να στοχεύει σε συγκεκριμένα μέτρα που θα δίνουν μια πρόσθετη αξία, θα δημιουργούν πρόσθετη αξία ως κέρδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως όφελος. Αυτό είναι ένα σημείο που πάντα τα κράτη-μέλη υπογράμμιζαν σε αυτές τις διμερείς επαφές που είχαμε κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου. Τώρα, κάτι άλλο οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι η καταπολέμηση των εγκλημάτων είναι κάτι το πολύ σημαντικό ως ε, υπόθεση. Αναμένουν οι πολίτες η συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγήσει στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της διασυνοριακή εγκληματικότητα και αναμένουν οι πολίτες ταυτόχρονα ελευθερία που θα διασφαλίζεται και δικαιοσύνη που θα εγγυόμεθα. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ασφάλειας που θα κατοχυρώνει τις άλλε πτυχέ. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αποβαίνει ει βάρο των ατόμων, των ε, πολιτών και πρέπει να είναι η ιδιωτική ζωή. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, μια αναλογία μεταξύ αυτών των μέτρων. Μέτρων προ όφελο τη ασφάλεια και μέτρων για τα δικαιώματα και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Όταν πρόκειται για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματο, οι προκλήσει είναι πάρα πολύ μεγάλε σίγουρα. Εμπόριο ναρκωτικών, εμπόριο ανθρώπων, τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων. Όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σίγουρα. Και ταυτόχρονα νέε μορφέ εγκλήματο προστίθενται σε όλε αυτέ τι γνωστέ ήδη μέσω του διαδικτύου, του ίντερνετ. Όταν πρόκειται για θέματα εγκληματικότητα, στην ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ολόκληρη σειρά αδικημάτων ή εγκλημάτων αναφέρονται, που είναι πιλωτικά, ας το πω έτσι, διάφοροι τομείς όπου διάφορες ιδέες και μεθόδους μεθοδολογικά θέλουμε να δοκιμάσουμε στον τομέα καταπολέμησης του εγκλήματος και στην εγκληματολογία καταπολέμηση ναρκοεμπορίου, καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων, καταπολέμηση κακοποίησης και εμπορίας παιδιών, ηλεκτρονικό έγκλημα στο διαδίκτυο, οικονομικά αδικήματα και εγκλήματα, διαφθορά. Όλα αυτά είναι αδικήματα ή εγκλήματα που απαιτούν μια συνεργασία για να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανευρωπαϊκή συνεργασία. Είναι πολύ θετικό το ότι εδώ επικεντρωνόμαστε και συμφωνούμε για αυτές τις προτεραιότητες. Το οργανωμένο έγκλημα λοιπόν στην Ευρώπη δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα σύνορα, ούτε σταματά εκεί. Και γι' αυτό θα πρέπει εμείς από πλευράς μας να δρούμε με τέτοιο τρόπο ώστε διασυνοριακά να καταπολεμούμε το έγκλημα. Να μην αποτελούν τα σύνορα πρόσκομα ή εμπόδιο για την καταπολέμηση των διασυνοριακών εγκλημάτων. Μια καλύτερη συνεργασία έχουμε ήδη διασφαλίσει στο επίπεδο των αρχών, των διοικητικών αρχών. Πρέπει πολλά περισσότερα να κάνουμε για να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική συνεργασία στον ποινικό τομέα από πλευρά μα και για την δίωξη των εγκλημάτων. Χρειαζόμαστε κοινή συνεργασία και μια καλά ανεπτυγμένη και ε, διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών κρατών των κρατών μελών, ένα αποτελεσματικό μέσο ανταλλαγής πληροφοριών και σίγουρα μια ανταλλαγή μεθόδων εργασίας μεθοδολογικά είναι σημαντικά θεμέλια και πρέπει να δούμε και τη λειτουργική συνεργασία. Για τη λειτουργική συνεργασία, λειτουργούσα συνεργασία, οι διάφορες αντιπροσωπείες διμερώς στις συζητήσεις που είχαμε εξέφρασαν ότι επιθυμούν να υποστηρίξουν περισσότερο την Ευρωπόλ και βλέπουν ότι πρέπει να έχει η Ευρωπόλ ένα σημαντικό ρόλο. Η Ευρωπόλ είναι ένα σημαντικό εργαλείο, ένα σημαντικό μέσο ώστε να με τη συνεργασία μας στην καταπολέμηση διασυνοριακών εγκληματικών πράξεων. Μπορεί να είναι ένα κομβικό σημείο για τη συνεργασία των ευρωπαϊκών διοκτικών αρχών, αστυνομικών αρχών. Αλλά μπορεί επίσης και στο διεθνές επίπεδο να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να πρέπει να ενταθεί αυτή η συνεργασία. Μια έκτακτη συνάντηση υπουργών στη Χάγη θα διεξαχθεί ε, τον Οκτώβριο ώστε να συζητήσουμε το μελλοντικό ρόλο της Ευρωπόλ. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής Λίμπε προσκαλείται φυσικά, είναι αυτονόητο αυτό, σε αυτή τη συνεδρίαση εκεί τότε. Ένα σημαντικό τμήμα ένα σημαντικό τμήμα της αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας σε αυτά τα επίπεδα είναι για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και της εγκληματικότητα, έγκυται και σε ένα, σε ένα καλό σύστημα ανταλλαγών πληροφοριών αμοιβαία. Οι εθνικές αστυνομικέ αρχές έχουν πληροφορίες εδώ που μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Αυτό γίνεται ήδη στο πλαίσιο της ε, νομικής ε, ε, για νομικά θέματα συνεργασίας και πρέπει να επεκταθεί και να τυποποιηθεί ως συνεργασία ώστε η ανταλλαγή πληροφοριών συνολικά να είναι πιο αποτελεσματική μεταξύ των αρχών. Είναι σημαντικό λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι σε αυτές τις ανταλλαγές πληροφοριών κύρια θεμελιώδη αιτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα λαμβάνονται υπόψη και ότι δεν θα, δεν θα διατίθενται περισσότερες πληροφορίες από ότι είναι αναγκαίο και ούτε θα αποθηκεύονται περισσότερες πληροφορίες για προσωπικά δεδομένα από, ότι είναι αναγκαίο. Θέλουμε να είναι μια ασφαλής περιοχή η Ευρώπη όπου θα καταπολεμάται το οργανωμένο έγκλημα όμως ταυτόχρονα πρέπει η ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα να προστατεύονται. Αυτή η εξίσωση μπορεί να λειτουργήσει και το ένα σκέλος να ικανοποιήσουμε και το άλλο. Μπορεί να γίνει αυτό. Στις διμερείς επαφές τώρα, πολλά κράτη-μέλη τι έκαναν. Υπογράμμισαν πολλά κράτη-μέλη πόσο σημαντικό σημαντικό είναι το θέμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα, νομικά, τα, θέματα ε, νομικών πλαισίων, διατάξεων και διεργασιών. Είναι αποφασιστική σημασία η αμοιβαία εμπιστοσύνη για να λειτουργήσει σωστά η συνεργασία μας. Πρόκειται για αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των εθνικών μας αρχών, αλλά και για την εμπιστοσύνη των πολιτών από την άλλη πλευρά, στα μέτρα που αποφασίζουμε και υιοθετούμε. Τα οι αρχέ των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται η μία στην άλλη, ώστε οι αμοιβέ αποφάσει και ε, να λαμβάνονται υπόψη και να είναι αποτελεσματικέ, να είναι σεβαστέ και αποτελεσματικέ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανήκουν μέτρα όπως κατάρτιση, εκπαίδευση, προγράμματα επιμόρφωση κατάρτισης και εκπαίδευση, όπω τα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εδώ υπόψη να δημιουργηθεί ένα είδο ανταλλαγών τύπου έρασμος, όσον αφορά τη, τους αστυνομικούς, τις διοκτικές αρχές. Και το, το πιο σημαντικό μέτρο για την ανάπτυξη αύξηση της εμπιστοσύνης είναι οι πολίτες να μπορέσουν να αποκτήσουν ελάχιστες προδιαγραφές που θα ισχύουν για δικαιοσύνη, για θέματα δικαιοσύνης. Άσχετα που θα ε, βρίσκονται και θα είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να είναι πολύ απλό αυτό και απλά να μπορεί να γίνει σε μια γλώσσα που θα είναι κατανοητή για αυτούς, να κατανοούν και να καταλαβαίνουν οι πολίτες γιατί κατηγορούνται για κάτι άσχετα αν είναι θύτες ή θύματα οι πολίτες και να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται σε δίκες. Είναι τουλάχιστον σημαντικό να υπάρξουν ελάχιστα δικαιώματα για τους εναγόμενους, για τους κατηγορουμένους σε ποινικέ διαδικασίες. Αν θέλουμε την ασφάλεια των πολιτών να την ενδυναμώσουμε, είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε τέτοια μέτρα που θα ενισχύουν την νομική βεβαιότητα, την νομική ασφάλεια και θα μπορέσουν να προαγάγουν τα δικαιώματα των πολιτών. Χρειαζόμαστε με άλλα λόγια εδώ ένα χρονοδιάγραμμα, ένα οδικό χάρτη, roadmap, για να γνωρίζουμε πώς θα, γίνει, πώς θα γίνουν όλα αυτά βήμα προς βήμα, σταδιακά και πρόκειται εδώ για συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα με στοχοθετημένες δράσεις και μέσα και εργαλεία που θα δημιουργούν πρόσθετη αξία για τους πολίτες μας. Ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν για παράδειγμα ένας κοινό μηχανισμός για την διερμηνία και μετάφραση για τα ποινικά θέματα. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει αυτό γοργά, σύντομα να υιοθετηθεί και να λειτουργήσει. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν τα θεμελιώδη δικαιώματα για εκείνους που θα είναι εναγόμενοι, κατηγορούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποινικέ διαδικασίες. Πρέπει όμως επίσης να διασφαλίσουμε και την προστασία των θυμάτων. Σίγουρα η ελευθερία κυκλοφορίας και ε, κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι οι πολίτες ταξιδεύουν πολύ περισσότερο περισσότερο και συχνότερα. Και έτσι είναι πολύ συχνότερα θύματα σε ένα κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο κατοικούν και είναι εγκατεστημένοι. Με άλλα λόγια, χρειάζονται προστασία, υποστήριξη, Πρέπει να συνδράμουμε αυτά τα άτομα, να έχουν πληροφορίες σε γλώσσα που είναι κατανοητή και εύληπτη για αυτούς. Χρειάζονται οι καταναλωτές επίσης βοήθεια και προστασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις ποινικέ αυτές δίκες και διεργασίες. Και πρέπει να διασφαλίζεται και ένα δίκαιο ποσό αποζημίωσης για αυτούς ως θύματα Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παλαιότερα θεώρησε σημαντική του προτεραιότητα και το υπογράμμισε. Ελπίζω λοιπόν να τύχω τη υποστήριξή σας και να έχουμε θετική επικοδομητική συνεργασία ώστε τα δικαιώματα των θυμάτων ποινικών πράξεων και αδικημάτων στην Ευρώπη να μπορέσουν να ενδυναμωθούν. Αυτά ήταν κάποια μερικά από τα πιο σημαντικά μείζωνα θέματα που απασχολούν την Σουηδία και άλλα κράτη-μέλη στη συζήτηση για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και έτσι υπογραμμίστηκαν. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω δύο λόγια ακόμα. Να πω ότι ελπίζω ότι θα έχουμε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών κατά το μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας και ευχαρίστω θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Καταρχήν όμως η συνάδελφή μου, η Υφυπουργό ε, Μίνα Γιούνκερ θα πει κάποια ε, λόγια για το θέμα του ασύλου και τα θέματα ενταξής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκράνερ. Κυρία Γιούνερ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ΛΥΜΠΕ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη ότι μπόρεσα να προσέλθω ενώπιον σας ως εκπρόσωπος της ε, Σουηδικής Προεδρίας ώστε να σας αναφέρω τα σχετικά με τις εξελίξεις και τις εργασίες για το πρόγραμμα, πρόγραμμά μας και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Πριν από ένα μήνα περίπου ε, οι υπουργοί μας και για τα θέματα μετανάστευσης ε, είχαν εμφανιστεί και για τα θέματα συνεργασίας και υπεγράμμισαν πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με την Ευρωβουλή για αυτά τα θέματα για Με τη σημερινή συνεδρίαση συνεχίζουμε ακριβώς σε αυτά τα οποία είχαμε προαναγγείλει. Από πλευρά ε, Υπουργού Μπίτστρομ ε, με αρμοδιότητα τα θέματα μετανάστευση, αναφέρθηκε πόσο σημαντικό είναι το ενδιαφέρον των πολιτών σε αυτά τα θέματα. Στην ε, Σουηδία συζητούμε ποια θα είναι η κατεύθυνση του προγράμματος της Στοκχόλμης. Αυτό γίνεται με παραδοσιακούς τρόπους, με blogs, με το διαδίκτυο, με το κατεστημένο και τις ομάδες του και με εκπροσώπους ε, ομάδων. Αυτό μας ικανοποιεί διότι αυτό είχαμε ακριβώς υπόψη το ε, ενδιαφέρον των πολιτών να μπορέσει να εκφραστεί και να βρεθεί στο επίκεντρο, να βρεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο των εργασιών για αυτό το πρόγραμμα. Δύο λόγια θα ήθελα να πω για τα θέματα μετανάστευσης, ε, χορήγησης ασύλου, ελευθερίας κυκλοφορίας μόλις ακούσαμε πιο πριν από τον Υφυπουργό ότι ένα από τα σημαντικότερα έργα της Σουηδικής Προεδρίας έγκυται ακριβώς στο να υπάρξει ένα νέο στρατηγικό πρόγραμμα για τον χώρο ελευθερίας, δικαίου και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά, θα έλεγα, έγγραφα που για αυτόν τον τομέα τα επόμενα χρόνια θα συνταχθούν και θα είναι διαθέσιμα και θα δείχνει κατευθύνσεις προς το μέλλον. Εμείς τι στοχεύουμε. Στοχεύουμε να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα με το οποίο θα δημιουργήσουμε μια πιο ασφαλή και πιο ανοιχτή Ευρώπη και θα οικοδομήσουμε μια πιο ανοιχτή και ασφαλή Ευρώπη όπου θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα των πολιτών. Στον τομέα μετανάστευσης και θεμάτων ασύλου Κατά τα τελευταία έτη έγιναν πάρα πολλά πράγματα, οπωσδήποτε. Ελήφθησαν αποφάσεις για το κοινό νομοθετικό πρόγραμμα. Ε, πρώτα βήματα έγιναν για μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ένα κοινό ε, σύστημα που θα διέπει τα θέματα ασύλου. Τα περισσότερα μέτρα τα οποία στο πρόγραμμα της Χάγης ε, εμπεριέχονται έχουν εκτελεστεί ή ευρίσκονται υπό εκτέλεση τώρα. Και αυτό είναι κάτι που μας ικανοποιεί σίγουρα ιδιαίτερα. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2004 σε, αυτή την πρόοδο που σημειώθηκε διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Σημαντικός λοιπόν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πέρα από αυτά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πέρυσι έκανε ε, προέβη στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Με βοήθεια αυτής της συμφωνίας, αυτού του συμφώνου, τα κράτη-μέλη υποχρεώθηκαν, ανέλαβαν την δέσμευση να εργαστούν για μια δίκαιη, συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απορρέουν από θέματα μεταναστευτικά, από την ίδια τη μετανάστευση και σε σχέση με τα θέματα ασύλου. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια ας το πω έτσι, ισχυρή πολιτική δύναμη που δημιουργήθηκε σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το επίπεδο. Θέλω όμως να πω ότι με αυτό το σύμφωνο δεν είπαμε και την τελευταία λέξη. Δεν είναι η τελευταία λέξη. Είναι βάση, αφετηρία, θεμέλιο για την περαιτέρω εργασία. Μία ολόκληρη σειρά διαβουλεύσεων θα υπάρξουν με τα εθνικά κοινοβούλια για παράδειγμα και έχουν γίνει ήδη κάποιες τέτοιες επαφές με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, με ε, εκπροσώπους εθελοντών, με εκπροσώπους πολιτών, με την κοινωνία των πολιτών. Τώρα η δουλειά αυτή που έγινε στο παρελθόν πρέπει να επικεντρωθεί σε δέσμες, σε συγκεκριμένα στοχοθετημένα μέτρα, με πάντα έχοντας υπόψη τη μελλοντική προοπτική, το μέλλον. Μια πολύ σημαντική συνεισφορά είναι η ανακοίνωση της Επιτροπής ε, για τα θέματα της ασφάλειας και δικαίου. Είναι η ανακοίνωση του Ιουνίου. Αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Στοκχόλμη συζητήθηκε τον Ιούλιο. Και είναι και η δική μου εντύπωση προσωπικά ότι έχουμε μεγάλη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των κρατών μελών. Επιτυγχάνεται ευρύτερη συμφωνία όταν πρόκειται για τις κατευθυντήριες γραμμές που αποτελούν, εμπεριέχονται σε αυτή την ανακοίνωση και αποτελούν τμήμα της. Ένα σημαντικό σημείο ως αφετηρία σε αυτήν την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακριβώς το σημείο που αφορά την καλή διαχείριση των θεμάτων μετανάστευσης. Αυτό αναφέρθηκε και στην Υπουργική Συνάντηση στη Στοκχόλμη. Αυτό για όλους μας έχει μεγάλη σημασία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά αλλά και για τα κράτη που είναι κράτη προέλευσης των μεταναστών και, όταν, και αν θέλουμε να τηρήσουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας και αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η πιο δυναμική, πιο ανταγωνιστική οικονομία παγκόσμια τότε θα πρέπει να ανοίξουμε την Ευρώπη για μια πιο ενδυναμωμένη μεταναστευτική πολιτική εργατικού δυναμικού από ό,τι συμβαίνει μέχρι σήμερα. Αυτό πρέπει να γίνει, διότι δεν πρέπει να αγνοήσουμε και τις δημογραφικές εξελίξεις, την υπεργύρανση της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε μια οικονομική κρίση. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και να προβληματιστούμε ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά τα επόμενα πέντε έτη, την επόμενη πενταετία και πέρα από αυτή την πενταετία το ε, μέλλον ως ευρύτερο ορίζοντα. Η οικονομική κατάσταση θα αλλάξει σε αυτό το μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να προτείνουμε αλλαγές, μεταρρυθμίσεις τώρα. Τώρα θα πρέπει να προταθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις που θα είναι αναγκαίες στο μέλλον. Τις χρειάζεται αυτές τις μεταρρυθμίσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξεύρει πρικισμένους εργαζόμενους με τα αναγκαία προσόντα, γιατί θα τους χρειαστεί αυτούς. Όταν λοιπόν θα έχουμε αυτά τα θέματα οικονομίας που θα έχει ανακάμψει, τότε θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις όσον αφορά το εργατικό δυναμικό. Με το πρόγραμμα προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις σε διαφορετικά ερωτήματα. Και αυτό ως προς το ότι θετικές επιπτώσεις της μετανάστευσης θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν και να βελτιστοποιηθούν και για τις κοινωνικές εξελίξεις, για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τρίτα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα συμβαίνει το ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν πόσοι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν και πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην αγορά εργασίας τους και στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει από κοινού με συντονισμένο τρόπο <clears throat> να καταπολεμήσουν την παράνομη ανεργία. Υπάρχει συμφωνία γι' αυτό, σίγουρα. Η πολιτική επιστροφής, παλινόστησης, η επαναπροώθηση παράνομων μεταναστών είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα, ένα αναγκαίο ε, στοιχείο για την αξιοπιστία της μεταναστευτικής μας πολιτικής. Εδώ η Frontex διαδραματίζει ένα πολύ αποφασιστικό ρόλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κράτη-μέλη επιθυμούν και θα ενισχύσουν αυτή την ε, υπηρεσία και την ε, διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Η ενίσχυση της Frontex όμως είναι ένα μέσο μεταξύ πολλών άλλων μία δράση μεταξύ πολλών άλλων. Μία ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών προέλευσης και των χωρών διαμετακόμισης, χωρών διέλευσης, είναι πολύ αναγκαία στοιχεία. Η αναπτυξιακή συνεργασία με αυτές τις χώρες πρέπει να ενταθεί, ώστε η ασφάλεια, η σταθερότητα και η μακροπρόθεσμη αηφορία, η βιωσιμότητα να διασφαλιστεί. Στην καταπολέμηση της παράνομης ανεργίας, ε, μετανάστευσης, με συγχωρείτε, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αναγκαία ισορροπία, ώστε τα μέτρα ασφάλειας να μην αποβούν εις βάρος της νόμιμης μετανάστευσης, των νόμιμων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή <clears throat> με το ότι η πρόσβαση στα θέματα ασύλου θα δυσχερανθεί για τους ετούντες άσυλο ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν ευαίσθητες ευπαθείς ομάδες όπως παιδιά ασυνόδευτα που ταξιδεύουν μόνα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αντιμετωπιστεί. Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης λοιπόν πρέπει να εμπεριέχονται εκείνα τα στοιχεία ακριβώς με τα οποία θα καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση και θα ελεγχθεί και θα αναχαιτιστεί και ταυτόχρονα όμως θα διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των, της προστασίας των όσων έχουν ανάγκη. Εδώ και θέματα αλληλεγγύης και επιμερισμού βαρών πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έγινε λόγος για αυτά. Πολλά κράτη ιδιαίτερα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη πίεση και τριβές από θέματα μετανάστευσης. Είναι μεγάλη πρόκληση για μας και πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα κράτη. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη σφαιρική προσέγγιση, μακροπρόθεσμα και χρειαζόμαστε διαφορετικής φύσεως μέτρα για να δράσουμε αποτελεσματικά. Πρέπει να δούμε σε σχέση με τα σφαιρικά θέματα μετανάστευσης και εξειδικευμένες προτάσεις από την άλλη πλευρά προτάσεις που θα αφορούν την πολιτική επιστροφής παράνομων μεταναστών, επαναπροώθησής τους ε, στις ε, χώρες διαμετακόμισης ή στις χώρες προέλευσής τους. Με τη Μάλτα βρισκόμαστε σε επαφές για ένα πιλωτικό σχέδιο και για άτομα τα οποία ε, την χάνουν προστασίας από την πείρα αυτού του πιλωτικού προγράμματος θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Το, ο στόχος μας ποιος είναι, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μα χειροπιαστά έναντι των κρατών μελών και έναντι τρίτων κρατών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις ή τριβές λόγω μετανάστευσης ή που τα συστήματα παροχής ασύλου επιβαρύνονται ιδιαίτερα από τους ετούντε άσυλο Επιπλέον έχουμε τον στόχο ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου που θέλουμε να δημιουργηθεί και να διευρυνθεί. Αφετηρία πρέπει να είναι ότι ο ετών άσυλο πρέπει με τα ίδια κριτήρια να αντιμετωπίζεται και να κρίνεται, να αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια. Άσχετα σε ποιο κράτος μέλος θα θέτει την αίτησή του, θα υποβάλει αίτηση για άσυλο και άσχετα σε ποιο κράτος μέλος θα ε, καταλήγει πρώτα από όλα τα κράτη-μέλη και κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα αυτό και το κοινό σύστημα ασύλου πρέπει να διευρυνθεί, να αποκτήσει σάρκα και οστά και να είναι αποτελεσματικό και να είναι ένα κοινό σύστημα και από κοινού να αποφασιστεί και να εγκριθεί. Αυτή λοιπόν η πρακτική συνεργασία θα πρέπει να βελτιωθεί καλύτερα και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να πετύχουμε το στόχο μας μέσα από αυτές τις βελτιώσεις. Μία άλλη πτυχή του κοινού συστήματος ασύλου είναι η εξωτερική διάσταση. Με την εξωτερική διάσταση έχω υπόψη εδώ την εγκατάσταση ε, προσφύγων και θέματα εγκατάστασης στα κράτη-μέλη προσφύγων από τρίτες χώρες. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται προστασία αλλά που δεν καταλήγουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πάνε σε άλλες ασφαλείς χώρες. Πρόκειται για ανθρώπους που έμειναν κάποτε κάπου σε ένα στρατόπεδο προσφύγων και δεν μπορούν ε, να προστατευθούν και δεν έχουν επιρροή στα θέματα προστασίας τους. Από κοινού λοιπόν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να πράξουν πολλά για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Μέσω μετεγκατάστασης για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα υπέβαλε μια πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα αυτά που χρήζουν προστασίας. Και μια σειρά κρατών μελών θα ήθελαν να ενταχθεί αυτό το σημείο, να εμπεριέχεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Η Σουηδική Προεδρία ελπίζει ότι κατά τη διάρκεια των φθινοπορεινών μηνών θα υπάρξει στενότερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, ώστε το πρόγραμμα για την επανεγκατάσταση ή μετεγκατάσταση αυτών των ατόμων γοργά να μπορέσει να εκτελεστεί. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Όπως και ο Υφυπουργός προανέφερε, εμείς το Σεπτέμβριο είχαμε διαφορετικού εκπροσώπου των κρατών μελών που προσήλθαν στην Στοκχόλμη, τους συναντήσαμε και συζητήσαμε συζητήσαμε μαζί τους αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτές τις συζητήσεις και διμερείς επαφές ε, τα κράτη-μέλη εξέφρασαν και συμπλήρωσαν με τις απόψεις τους αυτά που οι υπουργοί τους είχαν συζητήσει ήδη τον Ιούλιο προηγούμενα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατέστη σαφές, αποσαφηνίστηκε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της αποτίμησης, της αξιολόγησης των μηχανισμών αυτών των προγραμμάτων, ώστε να καταλάβουμε και να δούμε καλύτερα ποιες ανάγκες υπάρχουν και ποιες νέες προτάσεις πρέπει να υποβληθούν. Πρέπει κάπως να στρέψουμε το, το βλέμμα προς τα πίσω, στο παρελθόν, αλλά και για να μπορέσουμε να πορευτούμε σωστά προς το μέλλον και να κάνουμε αυτό που είναι αναγκαίο. Το δυναμικό μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από πλευρά χωρών χωρών λοιπόν, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εντυπωσιακά έχει υπογραμμιστεί σε πολλές παρεμβάσεις. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ε, για θέματα ασύλου θεωρήθηκε και αυτό μια σημαντική πρωτοβουλία, ένα σημαντικό στοιχείο. Η σημασία που έχει η ολοκλήρωση και η ένταξη όλων αυτών των θεμάτων ε, όσον αφορά και την εξωτερική διάσταση στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που υπογραμμίστηκε. Στη συνέχεια μετά από αυτές τις συζητήσεις και μετά από την άτυπη συνάντηση των Υπουργών στη Στοκχόλμη Τώρα πλέον εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης να πάρει σάρκα και οστά και να μπορέσει να επεκταθεί, να ε, λειτουργήσει σωστά. Ελπίζουμε ότι θα αποσαφινιστούν οι προτεραιότητες και ότι θα αντανακλώνται σε αυτές τις προτεραιότητες οι ανάγκες των πολιτών μας χρειαζόμαστε και επιθυμούμε μια ανοιχτή, διαφανή διαδικασία όπου όλα τα κράτη-μέλη, ε, τα θεσμικά όργανα και όσοι θα εμπλέκονται θα έχουν ε, σημαντικό ρόλο. Πρόκειται για ομαδική δουλειά, ομαδικό έργο και όχι ατομικό. Και λέω ότι κατά τη διάρκεια των ε, μηνών του φθινοπόρου θα έχουμε μια ολόκληρη σειρά επικοδομητικών επαφών και συζητήσεων με την Ευρωβουλή. Η συνεργασία σας είναι πολύ σημαντική για μας για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Στο τέλος τέλος Χρειαζόμαστε ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί να μα εκπροσωπεί και να το κάνουμε δεκτό όλοι. Και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Είμαι στη διάθεσή σας με χαρά να απαντήσω ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λούγκρεν. Γνωρίζουμε όλοι ότι το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις δραστηριότητες επιτροπής μας εφόσον βέβαια εγκριθεί και η συνθήκη της Λισαβόνας. 20 συνάδελφοι που να πάρουν το λόγο. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας παρακαλώ να περιοριστείτε σε παρεμβάσεις δύο λεπτών το μέγιστο. Ο κύριος Μπουζουτήλ πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους δύο ομιλητές ε, για τις ενδιαφέρουσες ε, τοποθετήσεις σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Εγώ θέλω να σταθώ στην κοινή πολιτική για την μετανάστευση και το άσυλο και να σας πω τα εξή. Βέβαια, θέλω να πω, ποιο είναι ο πολιτικός μας στόχος σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να είναι σαφής ο πολιτικός μας στόχος διότι θα πρέπει να αποκτήσουμε μία κοινή πολιτική για τη μετανάστευση και για το άσυλο που να είναι και δίκαιη αλλά και ισχυρή. Τι θέλει να πει δίκαιη. Δίκαιη για αυτούς που είναι δικαιούχοι της προστασίας. Δίκαιη έναντι των χωρών εκείνων οι οποίες δέχονται ένα, μια, ένα δυσανάλογο άχθος από αυτήν τη μετανάστευση. Επίσης θα πρέπει να σεβαστούμε την ευρωπαϊκή επικράτεια και πρέπει να είμαστε αυστηροί έναντι αυτών που δεν δικαιούνται να κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να τους το πούμε καθαρά και εξάσπτερα ότι η επιλογή τους είναι να ξαναγυρίσουν πίσω στους τόπους τους. Εμείς ε, συμφωνούμε απόλυτα με την προτίμηση που δίνεται στην εκούσια επιστροφή Υπάρχουν πολλά σχέδια στις διάφορες χώρες για την εκούσια επιστροφή που λειτουργούν και θα πρέπει να τα ισχυροποιήσουμε αυτά τα σχέδια διότι είναι πολύ πιο εύκολο να επαναπατριστεί κάποιος ε, εκούσια και όχι με το ζόρι. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται περισσότερη συνεργασία. Συνεργασία για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να διαπιστώσουν πώς έχει κατάσταση και να οργανώσουν κοινά ταξίδια επαναπατρισμού. Γνωρίζουμε ότι χωρίς την συνεργασία των τρίτων χωρών δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε τίποτα και για τις τρίτε χώρες αναφέρομαι ανοιχτά στη Λιβύη και στην Τουρκία που πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους στη διεθνή συνεργασία. Θα πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι αυτές οι χώρες έχουν πρόβλημα οι ίδιες για την προστασία των εξωτερικών τους συνόρων. Άρα και εμείς θα πρέπει να τους βοηθήσουμε ούτω ώστε να φυλάσσουν με καλύτερο τρόπο τα εξωτερικά του σύνορα. Η σύμβαση της ε, Γενέβης ε, πρέπει να γίνεται σεβαστή. Χρειάζεται ένα γραφείο της ε, συμπατίας των προσφύγων που να εργάζεται σωστά και χρειαζόμαστε επίσης και εγκαταστάσεις που να μπορούν να προσφέρουν παραπάνω πράγματα στις τρίτες χώρες για το Frontex. Θα πρέπει να εξετάσουμε τι έχουν κάνει οι τρίτες χώρες οι οποίες δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους ή το επίπεδο συμμετοχής ήταν χαμηλό. Επίσης, σχετικά με το θέμα της αλληλεγγύης. Και εδώ ολοκληρώνω. Ασκούνται πολλές πιέσεις. Να είστε σύντομος λέει ο πρόεδρος. Μία κουβέντα μόνο κύριε πρόεδρε. Έλεγα λοιπόν στις χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι αυταπάγγελτα θα πρέπει να σώζουν και να υποδέχονται όλους ε, όσους έρχονται και δεν μπορούν να επαναπατριστούν. Διαμορφώνεται λοιπόν η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι οι χώρες του Νότου από μόνες τους θα πρέπει να υποδεχθούν όλον αυτόν τον κόσμο. Μα δεν είναι αυτό το πράγμα αλληλεγγύη. Αν θέλουμε εμείς να μιλήσουμε για αλληλεγγύη θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε όλα αυτά να είναι αποτελεσματικά. Σας... Δύο λεπτά έχετε, ούτε τέσσερα ούτε πέντε, δύο. Διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε στο χρόνο που έχουμε. Τουλάχιστον 20 μέλη ζήτησαν να παρέμουν και σήκωσαν το χέρι τους. Αν δεν τηρήσετε αυτό το χρονικό όριο δεν θα φτάσει ο χρόνος. Η κυρία Χάνης Πλέσχατ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πανσύντομη. Ο Υπουργός είπε ότι η αφετηρία για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου. Ε, εμείς έχουμε ένα φύλλο πορείας σχετικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται στα κράτη-μέλη αλλά το οποίο δεν λειτουργεί γιατί το Συμβούλιο δεν αποφασίζει. Εγώ έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη και εκτιμώ ιδιαίτερα τις φιλοδοξίες σας αλλά αυτό δεν φτάνει για να πείσει τους αρχηγούς κρατών κρατών και κυβερνήσεων. Πρέπει να περάσουμε στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία και για την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης θα είμαι σύντομη. Μα φυσικά και εδώ υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Δεν υπάρχει συμφωνία σε τελευταία ανάλυση για την προστασία των συνόρων, για την... Ε, κοινή χορήγηση ασύλου για όσους θα πρέπει να εκδιωχθούν, ε, για όσους ε, ε, θα πρέπει να βοηθηθούν. Μιλάμε για αλληλεγγύη σε όλους αυτούς τους τομείς. Μα πότε όμως θα υπάρξει κάτι το συγκεκριμένο μέσα σε όλα αυτά, διότι όλα είναι πάρα πολύ ωραία στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Όλοι θα θέλαμε να, να, να ήταν πραγματικότητα, αλλά ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα θέσαμε ένα όριο το 2010 και πάλι φεύγουμε από αυτό το όριο. Το παρατείνουμε. Για τα, για τα θεμελιώδη δικαίωμα ο Προεδρεύων του Συμβουλίου μίλησε για ίσα δικαιώματα για όλους. Εγώ έθεσα ε, για την ε, Λετωνία ε, γραπτές ερωτήσεις στο Συμβούλιο και κανένας δεν μου απάντησε και μου είπανε μάλιστα σήμερα το πρωί ότι το Συμβούλιο δεν τις είδε καν. Μα αυτό είναι σκανδαλώδες. Το Συμβούλιο θα πρέπει να διορθώνει όλες αυτές τις καταχρηστικές καταστάσεις. Πρέπει να μιλάει όταν κάτι δεν δουλεύει στην Ευρώπη, κάτι δεν λειτουργεί. Το ίδιο πρέπει να κάνει και για τις ποσοστώσεις του γάλακτος, και τα ίδια και για τη Ρωσία και για την παραβίαση φυσικά των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Θα το προσπαθήσω, Πρόεδρε όπου κρίμα είναι ότι μόνο τόσο λίγο χρόνο έχουμε ώστε πραγματικά βουλευτές που έχουν ασχοληθεί σε βάθος με το πρόγραμμα της Στοχόλμης να αναγκάζονται να είναι τόσο σύντομοι. Αυτό είναι κρίμα. Λοιπόν, Κάπως επιφανειακά θα μείνω στην επιφάνεια παρόλα αυτά. Ευχαριστώ τους υφυπουργούς, τον υφυπουργό για την παρουσίαση και για τη βούληση η ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών να, είναι επίκεντρο των προσπαθειών μας και στον τομέα των προσωπικών δεδομένων και της προστασίας τους. Τρία σημεία θέλω να θέσω στο επίκεντρο. Αφενός το γεγονός ότι στο πρόγραμμα, όπως εγώ το διάβασα μέχρι τώρα, εξακολουθεί ο τομέας αυτής της ενίσχυσης να μην είναι γενικός, σε ένα γενικό επίπεδο. Λείπουν οι εξειδικευμένε προσεγγίσεις και στον τομέα της αξιολόγησης, αποτίμηση, τα υφιστάμενα μέτρα α το πω έτσι, δεν είναι πολύ συγκεκριμένα ή εξειδικευμένα. Και εδώ έχει πει και το Σουηδικό Κοινοβούλιο με σαφήνεια ότι μια πλήρης αξιολόγηση πρέπει να γίνει πριν από την υιοθέτηση νέων μέτρων για την ασφάλεια και νέων μέτρων για την επιτήρηση και εποπτεία. Αυτά είναι απόλυτα αναγκαία και σημαντικά στοιχεία ως παρατηρήσεις ώστε σε σχέση με την πρόληψη να επικεντρωθούμε σε αυτήν και όχι στην καταστολή και καταδίωξη. Και όταν έχουμε γενικές υποψίες και όχι εξειδικευμένες υποψίες, ε, τότε οι πολίτες ε, αν δεν, υπάρχουν, αν δεν υπάρχει εξειδίκευση είναι κάτι που τους κάνει και υποφέρουν. Τώρα στην καταπολέμηση των εγκλημάτων δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί υποχρεωτικά με μεγαλύτερη εποπτεία και επιτήρηση ή καταστολή, αλλά με ενίσχυση της πρόληψης και ενίσχυση των, της αστυνομικής συνεργασίας επιτόπου και όχι με ένταση των αστυνομικών μέτρων. Μια πραγματική πρόληψη δεν μπορεί να επιτευχθεί με εποπτεία, με επιτήρηση, με κάμερες κτλ. Και το πώς μπορεί να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της δίωξης ε, αφενός ε, και των μέτρων ασφάλειας και από την άλλη πλευρά της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ισόρροπη σχέση στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης για αυτά. Ευχαριστώ. Mr. τριανταφυλλίδη Κύριος Τριανταφυλλίδης παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Σουδικής Προεδρία και να αναφέρω ότι σε ό,τι αφορά την ομιλία της ε, κυρίας Λιούγκρεν στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες για δημιουργία γραφείου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Προερχόμενος από ένα κράτος μέλος όπως η Κύπρος, το οποίο έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο με δυσανάλογες αιτήσει ασύλου σε σχέση με τα κοινωνικά και οικονομικά του δεδομένα, λόγω κυρίως της γεωγραφικής του θέσης, των πολιτικών αλλά και δημογραφικών καταστάσεων, θεωρούμε πως η δημιουργία αυτού του γραφείου θα βοηθήσει σημαντικά στην επίλυση πολλών προβλημάτων, κυρίως ανθρωπιστικών, που αφορούν τη στήριξη των ατόμων που αιτούνται άσυλο, αλλά και στον καλύτερο συντονισμό. Είναι ένα μέτρο το οποίο προωθεί τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και από το οποίο θα επωφεληθούν σημαντικά οι μεσογειακές χώρες, οι οποίες είναι και οι κύριες χώρες υποδοχής των ετούντων ασύλου. Λόγω του προαναφερθέντος, πρέπει να τονίσω τη σημασία του να δημιουργηθεί αυτό το γραφείο σε κράτος μέλος της Μεσογείου. Αυτό θα βοηθήσει τους ειδικού να διεκπαιρεώσουν καλύτερα το έργο τους και να κατανοήσουν την ιδιόμορφη κατάσταση που δημιουργείται σε χώρες πρώτης γραμμής, που δέχονται τις περισσότερες αιτήσει ασύλου και χρησιμοποιώντας αυτή την εμπειρία να συνεισφέρουν καλύτερα στο όλο έργο της υπηρεσίας υποστήριξης για το άσυλο. Γνωρίζοντας τη σημασία του έργου που μπορεί να επιτελέσει αυτό το γραφείο, Τονίζω καλά, ε, ξανά κύριε Πρόεδρε και κλείνω την ανάγκη δημιουργίας του το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε κυρία Κέλλε. Σας ευχαριστώ. Έχω ένα πρόβλημα με τον όρο ισορροπία που χρησιμοποιήθηκε γιατί από τη στιγμή που μιλάμε για θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να ισχύουν παντού και για όλους κατά τον ίδιο τρόπο, κατά ένα ισορροπημένο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχετε λάβει κάποιες τροπολογίες από την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι ήταν σήμερα το πρωί μαζί μας. Θα ήθελα να εξετάσετε τις προτάσεις αυτές και θα ήθελα να γνωρίσω αν θα τις λάβετε υπόψη σας. Πρόκειται για μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, ασχολείται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι προφανές ότι οι προτάσεις τους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ε, περαιτέρω σύνταξη του προγράμματος της Στοκχόλμης. Και κάτι ακόμα. Συμφωνώ με τα όσα είπε η Υπηρεσία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης δικαιώματα αναγνωρίζονται μόνο για τους πολίτες. Τι γίνεται για αυτούς που δεν έχουν την ευρωπαϊκή υπηκότητα όμως. Αυτοί δεν αναφέρονται πουθενά και επομένως για αυτούς δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τα δικαιώματά τους. Και ξέρετε ότι υπάρχουν και ευρωπαϊκέ υπηρεσίε όπω η Frontex, οι οποίε έχουν εμπλακεί σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα σε βάλτε ομάδε όπω είναι οι μετανάστε. Και περαιτέρω η αξιοπιστία μα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να απορρέει μόνο από την από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι από την αποτελεσματικότητα μιας πολιτικής επιστροφής ή μετεγκατάστασης ε, κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να εξασφαλιστεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι με περισσότερη λεγγύη και με καλύτερη πολιτική για το άσυλο θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε πολύ θετικότερα αποτελέσματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη στιγμή που μιλάμε για εθελούσια μόνο αλληλεγγύη, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η αλληλεγγύη αυτή θα υφίσταται σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν χώρες ουσιαστικά που δεν παρέχουν τον, το απαραίτητο επίπεδο προστασίας προς ε, τους ετούντες άσυλο ακριβώς επειδή η αλληλεγγύη η οποία ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθαρά ε, εθελοντική, εθελούσια. Εγώ ήθελα να αρχίσω λέγοντας ε, στην Σουηδική Προεδρία ότι η Ευρώπη ούτως οικοδομείται σε αυτή τη φάση λοιπόν που οικοδομούμε την Ευρώπη, η Σουηδική Προεδρία δίνει το παράδειγμα για το πώς επιλύνονται τα προβλήματα τα οποία αφορούν στους Ευρωπαίους. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν τα εξή. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τη συμπεριφορά της Eurojust. Υπάρχει Επίσης το Συμβούλιο μία διαπίστωση ότι η εγκληματικότητα αποκτά έναν διεθνιστικό χαρακτήρα. Αρχίζει κανείς να σκέφτεται ποινικέ διώξεις σε ενιαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή πώς μπορεί να φανταστεί κανείς ας πούμε ότι για ένα αδίκημα υπάρχουν διαφορετικές, αν θέλετε και ανταγωνιστικές ποινές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η πορνεία τιμωρείται διαφορετικά από τη μία χώρα στην άλλη. Πώς το βλέπετε λοιπόν εσείς αυτό για, την, για μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση των διαφόρων αδικημάτων και πώς φαντάζεστε εσείς αντίστοιχα με το στο, θέμα του ασύλου ε, να αντιμετωπίσετε το θέμα των των ασυνόδευτων αντιλήκων, η κυρία Έμβελτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Σουηδικής Προεδρίας για την παρουσία τους στη συνεδρίασή μας. Η Σουηδική Προεδρία α, τα πηγαίνει πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να σταματήσουν τα επενετικά μου σχόλια. Ακούσαμε διάφορες παρεμβάσεις, ένθερμες θα έλεγα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, ότι επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στους πολίτες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα όλα αυτά. Δεν είμαι φύση κοινική, αλλά τελικά τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Όταν για παράδειγμα μιλάμε για την συλλογή προσωπικών δεδομένων, για την παρακολούθηση εποπτεία των πολιτών, θα ήθελα στην πράξη να γνωρίζω πού είναι τα όρια, πού τίθενται τα όρια, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν καθόλου όρια Κανένα περιορισμό, Ακόμα και η ίδια η Σουηδία έχει εγκρίνει δρακόντια μέτρα παρακολούθηση και εποπτείας των πολιτών. Ακόμα και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ελέγχουν. Δεδομένα DNA, σε ποιον μιλάνε, πού ταξιδεύουν, με ποιον μιλάνε στο, τηλέφωνο, πόσα χρήματα έχουν στο τραπεζικό του λογαριασμό. Πού σταματάει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα σήμερα να μάθω πού έχετε θέσει τα όρια και εξ ονόματος Συμβουλίου. Κάθε φορά που μιλάτε πολύ θετικά για την καταπολέμηση των διακρίσεων, για την ισότητα και ούτε καθεξής, η βουλευτής που κάθεται δίπλα μου έχει δώσει πάρα πολύ καλά παραδείγματα για τις περιπτώσεις εκείνες που το Συμβούλιο μας λέει ότι δεν εμπλέκεται στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών μελών. με εμεί είχαμε την εντύπωση ότι θεμελιώδη δικαιώματα και ισότητα είναι κάτι το καθολικό. Αν λοιπόν δεν προστατεύετε τα προσωπικά δεδομένα, αν δεν προστατεύετε τα θεμελιώδη δικαιώματα, αν δεν καταπολεμείτε τις διακρίσεις, τότε τι ακριβώς κάνετε, σε τι αναφέρεστε κάθε φορά που λέτε ότι εστιάζεστε στον πολίτη. Θα ήθελα πραγματικά να καταλάβω. Ένα ακόμα παράδειγμα, απόφαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ένας υπήκος των Φιλιππίνων ύποπτος για τρομοκρατικές δράσεις ε, μπήκε σε μία blacklist, σε ένα μαύρο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την 18η τέτοια απόφαση του δικαστηρίου, η, σύμφωνα με την οποία η συμπερίληψη υπηκών κατά αυτόν τον τρόπο σε μαύρες λίστες είναι παράνομη. Πόσες δικαστικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν για να καταλάβει το Συμβούλιο ότι πρέπει να σεβαστεί το κράτος δικαίου. Θα ήθελα πραγματικά να γνωρίζω γιατί μιλάτε όταν μιλάτε για θεμελιώδη δικαιώματα, όταν μιλάτε για ποιότητα, όταν μιλάτε για κράτος δικαίου. Στην πράξη πείτε μου τι προτείνετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Μποργέτσιου. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, παν σύντομες ερωτήσεις. Από αυτά που άκουσα από τον υπεύθυνο για τα εσωτερικά θέματα και τη δικαιοσύνη, ακούσαμε να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο πολύ θετικό ε, για όσα αναλαμβάνει η Σουηδική Προεδρία στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Στοκχόλμης και που θέλει να προτείνει για ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξη πιο συγκεκριμένα στο θέμα του ασύλου. Θέλω όμως να ρωτήσω στους αντιπροσώπους της Σουηδίας αν από αυτήν την τόσο απομακρυσμένη περιοχή, τόσο τόσο μακριά από τη Μεσόγειο και από τις χώρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, ε, αν πραγματικά έχει μία ε, εικόνα, μία ουσιαστική πραγματική εικόνα για την μετανάστευση στις χώρες δηλαδή που γεννιούνται πραγματικά τα δράματα, τα δράματα ε, τα οποία έχουν ως γεννησιουργό αιτία τις εγκληματικές οργανώσεις που αποτελούν και τους βασικούς υπεύθυνους ε, για την ε, άφηξη των ε, μεταναστών από τις τρίτες χώρες σε άθλιες συνθήκες. Βλέπω ότι... Βλέπουμε εμείς μάλλον σε ποια χάλια φτάνουν οι μετανάστες όταν έρχονται στη δική μας επικράτεια αλλά μπορούμε πια να σταματήσουμε και αυτή την τροπή, αυτό το έσχος του 20ου αιώνα που είναι το, το εμπόριο ανθρώπινης σάρκας. Λοιπόν, μπορούμε εμείς να αρχίσουμε Βέβαια αυτό θέλει, να, ε, θέλει κάποιος να έχει ενόραση και συνήθως την ενόραση την έχει κάποιος όταν τα βλέπει τα πράγματα από μακριά και όχι από κοντά. Και μίλαγε προηγουμένως ο Κύπριος συνάδελφος. Μα χώρες σαν την Κύπρο, τη Μάλτα και τη δική μου που είναι μεσογειακές χώρες πολλές φορές υποχρεούνται να παρεμβαίνουν ασυντόνιστα με ανεπαρκή μέτρα. Μπορούμε εμείς πια να κόψουμε το κεφάλι της λερναίας ύδρας του τέρατος αυτού που ασκεί αυτήν την απίστευτη αντιανθρωπιστική δραστηριότητα που είναι η διακίνηση των λαθρομεταναστών. Ο κύριος Μπρόνς και σας υπενθυμίζω το όριο χρόνου, το χρονικό όριο μιλίες. Παρακαλώ να το σεβαστείτε. Κύριε Μπρόντς, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λούγκρεν είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερους μετανάστες για μια πιο δυναμική οικονομία. Και ουσιαστικά απευθύνθηκε κατά αυτόν τον τρόπο στα άτομα όχι σαν πραγματικούς ανθρώπους αλλά σαν μονάδες παραγωγής. Εγώ νομίζω ότι ε, τα πράγματα θα πρέπει να ισχύουν αντίστροφα, ότι το βάρος θα πρέπει να δίνεται στον ίδιο τον άνθρωπο. Η μετανάστευση έχει παραμορφώσει πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης, ανεπανόρθωτα θα έλεγα. Και αν δείτε πολλές δημοσκοπήσεις θα δείτε ότι οι πολίτες της Ευρώπης θέλουν να σταματήσει πλέον μετανάστευση, δεν θέλουν υπόσχεση αένα, αένα ονρών μετανάστευσης. Θα μιλήσω ξεκάθαρα σήμερα το απόγευμα προκειμένου όλοι να συντοποιήσουν και να κατανοήσουν τι θέλω να πω και αναφέρομαι σε όλους εδώ πέρα τους συναδέλφους που είναι παρόντες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τη συντομία σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ενοχλήθηκα πολύ από την ιδέα αυτή της οικονομικής αποτελεσματικότητας, δηλαδή να αποτελέσει αυτό την κινητήρια δύναμη στη μελλοντική κοινοτική μεταναστευτική πολιτική, Καθώς εξελίσσεται η πολιτική μετανάστευση στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες θα πρέπει να είναι οι βασικές αρχές της πολιτικής αυτής. Και η ερώτησή μου προς τη Σουηδική Προεδρία είναι ακόλουθη. Πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη αποτελεί, θα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη αρχή της πολιτικής μετανάστευσης, της κοινοτικής και πιστεύετε ότι θα πρέπει να εξεταστεί το γενικότερο ζήτημα της μετανάστευσης στα πλαίσια τα σωστά, δηλαδή τα οικονομικά και κοινωνικά πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, δηλαδή να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια της μετανάστευσης. Ουσιαστικά στο δικαίωμα ενός ανθρώπου να παραμείνει στη χώρα όπου διαμένει στη χώρα καταγωγής του. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για τους περισσότερους μετανάστες η μετάβαση σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γίνεται ελαφριά την καρδία. Πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους, αφήνουν πίσω τους την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, τις κοινότητές τους και αυτό οφείλεται ακριβώς στις πολύ άδικες οικονομικές πολιτικές που ακολουθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου για παράδειγμα και γενικότερα η ε, γενικότερη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση που υπάρχει στο εμπόριο και την οποία σπάζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο δεν μιλάμε για τα κυριαρχικά οικονομικά κυριαρχικά δικαιώματα του τρίτου κόσμου από το να φερόμαστε μόνο στις φιλελεύθερες αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για ποιο λόγο δεν μιλάμε περισσότερο για οικονομική δικαιοσύνη. Μια οικονομική δικαιοσύνη που θα επέτρεπε στι κοινότητε αυτέ να παραμείνουν αλόβητε, να μην αναγκαστούν να αποσυντήθενται, να μην αναγκάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι να εγκαταλείπουν τι οικογένειέ του προκειμένου να βρουν εργασία. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το κέντρο τη συζήτηση κάθε φορά που μιλάμε για μετανάστευση. Και κάτι ακόμα. Να αναφερθώ στο ζήτημα των νέων κρατών μελών, ιδίω στο δικό μου το κράτο, στην Ουγγαρία θα ήθελα να αναφερθώ, Ορισμένες από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται, θα έλεγα ότι γίνονται σχεδόν χώρες του τρίτου κόσμου. Ε, ε, ε, έχουν φτάσει σε απόλυτο σημείο ένδυας και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τελικά εξαιτία των προγραμμάτων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν προωθηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, από την Παγκόσμια Τράπεζα και από άλλου οργανισμού, συντομεύεται λέει ο Πρόεδρο, έχουμε καταλήξει να γίνουμε κι εμεί χώρε υπανάπτυκτε του τρίτου κόσμου και παράλληλα ευδοκιμεί μια τεράστια παράνομη ε, οικονομία ε, διακινητών ε, εμπόρων ανθρώπων κακοποιών ουσιαστικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθεί αυτό υπόψη στα πλαίσια του προγράμματο Στοχόλμη. Εστιαστείτε σε χώρε σαν την Ουγγαρία όπου τα φαινόμενα μετανάστευση είναι παρόμοια τα φαινόμενα που έχουμε σε χώρε του τρίτου κόσμου. Σα ευχαριστώ. Προαναγγέλλω uh, ότι κλείνει ο πίνακα αγοριτών όσων θα παρέμβουν και δεν θα προσθεθούν άλλοι. Σύπερ παρακαλώ κυρία Σύπερ δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα δύο σημεία να αναφέρω. Στο παρελθόν επανειλημμένα μας είπαν και ακούσαμε πόσο σημαντική είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς στην καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος κτλ. Αλλά αυτό φαίνεται ακριβώς να είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή λείπει αυτή, απουσιάζει αυτή η εμπιστοσύνη. Η εντύπωσή μου είναι ότι συχνά τα μέλη του Συμβουλίου είναι αυτονόητο ότι λαμβάνουν τις αποφάσεις ότι πρέπει λέει να είμαστε επιτυχείς, όμως τα ίδια μέλη του Συμβουλίου, οι Υπουργοί όταν γυρίζουν στα κράτη-μέλη, στις χώρες τους, στην υλοποίηση και ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων, για να το πω με κάθε επιφύλαξη, είναι διστακτική μάλλον και επιφυλακτική είσαστε σε θέση αυτή την θέση την οποία εκφράζω να την ε, απορρίψετε και να διαφωνήσετε με αυτήν τεκμηριωμένα δεύτερον χώρος ασφάλειας δικαιοσύνης και δικαίου. Θέλω εδώ να αναφέρω κάτι που λείπει. Ένα, ένας χώρος της ασφάλειας δικαίου. Αυτό είναι σημαντικό. Για πολίτες μας, πάρα πολλούς πολίτες, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή αν ο συνταξιούχο δεν παίρνω, δεν μου επιστρέφονται τα νοσήλια και τα, το κόστο για φάρμακα ή αν ω Ευρωπαίο σε ένα τύχημα εμπλέκομαι και δεν υπάρχει υποστήριξη, αυτό δείχνει ότι οι πολίτε ε, βρίσκονται όλο και πιο μακριά από την Ευρώπη που δεν είναι σε θέση να ρυθμίσει αυτέ τι μικρολεπτομέρειε. Ανήκουν αυτά τα θέματα στο πρόγραμμα τη Στοκχόλμη ή αποκλείονται από αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρομέρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να σταθώ στην ε, γραμμή, στην προβληματική των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, στον ιδιωτικό βίο και μιλάω πιο συγκεκριμένα για τα θέματα προσωπικής βίας, κυρίως βίας κατά των γυναικών. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τη Σουηδική Προεδρία αν σκέφτηκε να συμπεριλάβει πώς μπορεί να υπάρξει πρόληψη των αδικημάτων άσκησης βίας κατά των γυναικών. διότι ορισμένα κράτη ήδη έχουν λάβει μέτρα ούτως ώστε αυτός ο χώρος δικαιοσύνης ε, και ελευθερίας ε, και δικαιοσύνης να είναι ένας χώρος και για τις γυναίκες. Εδώ δεν μιλάμε για προστασία δεδομένων, μιλάμε για φυσική προστασία, για τη σωματική ακεραιότητα των γυναικών. Δηλαδή, μέτρα που να δημιουργούν κίνητρα ούτως ώστε οι γυναίκες να καταγγέλουν την κακομεταχείριση ή μέτρα, ας πούμε, η απομάκρυνση αυτού που ασκεί τη βία κατά των γυναικών. Στατιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή πληροφόρησης ε, στα θέματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί μία βασική προτεραιότητα για τη Σουηδική Προεδρία. Εδώ δεν πρόκειται μόνο για προστασία των γυναικών αλλά και αποφυγή των αδικημάτων αυτών που στην ιδιωτική σφαίρα παραβιάζουν το χώρο των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Κυρία Φλότρο, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η δυσκολία του να πείσουμε για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι τελικά ότι είχαμε δύο προγράμματα πριν από τη Στοκχόλμη, του Ταμπέρε και της Χάγης. Και άμα δούμε από κοντά πώς σήμερα ασκείται η πραγματική προστασία των ετούντων άσυλων στην Ευρώπη, ε, πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε να, αυτά τα δύο προγράμματα που πολύ σωστά εσείς επαναλαμβάνετε και που εγώ θα ήθελα να έχουμε ένα κοινό σύστημα, ένα κοινό καθεστώς ευρωπαϊκού ασύλου. Στην Ευρώπη σήμερα παρά αυτά τα δύο προγράμματα δεν υπάρχει τίποτα. Πρώτον, δύσκολο είναι να έρθει κανείς στην Ευρώπη. Όλοι το ξέρουν και όλοι το λένε. Αλλά πρέπει όμως να ληφθούν και τα πραγματικά μέτρα ούτως ώστε στις διάφορες επιχειρήσεις Frontex ή σε οποιασδήποτε θαλάσσιες επιχειρήσεις όλοι οι ενδυνάμοι ετούντες άσυλο να μπορούν και de facto και ουσιαστικά τη δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο πράγμα το οποίο δεν το έχουν σήμερα. Εγώ έρχομαι από το καλή... Εσείς ακούσατε τελευταία να μιλάμε για το Σαγκάτα και μάλιστα για την ε, ζούγκλα, ε, αυτό το στρατόπεδο το οποίο το διέλυσαν αυτή τη εβδομάδα. Μα δεν μιλάνε καν για άσυλο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να πάνε ούτε στη Μάλτα ούτε στην Ελλάδα. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ζητάνε άσυλο οι άνθρωποι. Λοιπόν, ε, για αυτούς τους λόγους εμείς λοιπόν θα πρέπει να ξαναδούμε τις συμφωνίες του Δουβλίνου οι οποίες τελικά είναι ένα εμπόδιο για το άσυλο στην Ευρώπη και αυτή η πολιτική ε, ε, επανόδου και επαναπατρισμού μα αυτή η, λογική κράτησης των μεταναστών και κυρίως των ανήλικων παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα Πρέπει εμεί να πάρουμε αυτά τα βασικά δικαιώματα και το περιεχόμενό τους δηλαδή και να δούμε ότι δεν προστατεύουν σήμερα κανέναν και να λάβουμε πραγματικά μέτρα ούτω ώστε να βοηθήσουν την κατάσταση. Και εγώ προσδοκώ από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης να προχωρήσει στα σοβαρά προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω τους Σουηδούς εκπροσώπους της Σουηδικής Προεδρίας. Να ευχαριστήσω για την προαγωγή των θεμάτων αυτών. Καλωσορίζω λέγω τους Σουηδούς εκπροσώπους και ευχαριστώ για την παρουσίαση του προγράμματος Σουηδικής Προεδρίας. Κάνετε λόγο για μια ευρεία στρατηγική για την προστασία των παιδιών. Έχω συγκεκριμένη πείρα που έχω αποκομίσει σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή λοιπόν. Τώρα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 κράτη-μέλη πλέον, είμαστε σαν μια οικογένεια δηλαδή και ζούμε την ε, εξέλιξη, το βίωμα των ε, μεικτών, ανάμεικτων οικογενειών. Αυτά είναι καλά. Όταν όμως χωρίζουν οι οικογένειες, τότε τα παιδιά είναι τα θύματα του διαζυγίου, του χωρισμού. Και πολύ συχνά τι γίνεται. Διαφορετικές οργανώσεις εμπλέκονται οι οργανισμοί σε αυτή τη διαδικασία και ακόμα και τα δικαστήρια δεν μπορούν να λάβουν τις πιο σωστές και αναγκαίες αποφάσεις. Δεν θεωρείτε ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών και την προστασία των παιδιών θα έπρεπε να εμπεριέχει ένα στοιχείο που θα επιτρέπει πρώτα και κύρια, κυρίαρχα να προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών αντί να βοηθά τους διαδίκους για την αντιμετώπιση των επιχειρημάτων τους. Δεν νομίζετε ότι χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων που θα επιτρέπει στα ε, θεσμικά όργανα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κατάσταση. Άλλο θέμα είναι η μετανάστευση και η νόμιμη ε, μετανάστευση. Εσείς κάνετε λόγο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και αναχέτησης της σημείωσής της. Δεν συμφωνώ ότι ο κύριος στόχος μας είναι να μειωθεί να μειωθούν, να ελέγξουμε τα στοιχεία ή τα αίτια τα οποία προωθούν την παράνομη μετανάστευση. Δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν είναι αυτό η πρωταρχική μας προτεραιότητα. Διότι ουσιαστικά η ερώτησή μου, η παρέμβαση αυτή δημιουργεί τεράστια ε, πίεση στην αγορά εργασίας. Και όταν γίνεται λόγος για την μείωση, την αναχέτηση παράνομης μετανάστευσης, πολύ καλό θα ήταν να είχαμε εξειδικευμένα, πολύ συγκεκριμένα, πραγματιστικά, ρεαλιστικά μέτρα και όχι λόγια. Η κυρία Έρντς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ με κάνει και προβληματίζομαι και με στενοχωρεί κάπως θα έλεγα αυτά που η Σουηδική Προεδρία ανέφερε για την πολιτική ασύλου. Νομίζω ότι ξεπερνά τις πραγματικές ανάγκες και τις παρακάμπτει κατά πολύ. Θέλετε να καταπολεμήσετε, είπατε το έγκλημα, την εγκληματικότητα. Θέλετε μεγαλύτερη ασφάλεια, λέτε. Η μόνη απάντηση που έχετε είναι η διασύνδεση των μέσων εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας και αμελείτε και είσαστε τυφλοί προς την ίδια την πραγματικότητα. Ποτέ δεν αξιολογήσατε την Frontex, ποτέ δεν ελέγξατε την ε, Frontex. Τώρα θέλετε να την μεγιστοποιήσετε και να την βελτιστοποιήσετε. Διερωτώ με τι γίνεται με την ασφάλεια εκείνων που βρίσκονται μπροστά στις πύλες, ε, στις πύλες της Ευρώπης και για κάθε εύλογο λόγο που έχουν θέλουν να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη. Αυτά τα ερωτήματα μένουν αναπάντητα. Θα ήθελα να μου πείτε, να μου απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτη, τι γίνεται σε σχέση με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Τι γίνεται ώστε λιγότεροι άνθρωποι να βρίσκονται ενώπιον των πυλών της Ευρώπης και να πεθαίνουν στις πύλες της Ευρώπης επειδή είναι ε, στεγανό αυτό το φρούριο Ευρώπη και δεν έχουν ευκαιρία να μπουν σε αυτό. Δεύτερο, αναφέρατε η παράνομη μετανάστευση πρέπει να καταπολεμηθεί λέει φτάνουμε σε τέτοιε έννοιες τώρα που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην αντιμετώπιση τους. Μπορεί κανείς πολύ γρήγορα από την νομιμότητα να καταλήξει στην παρανομία. Νομιμότητα και παρανομία βρίσκονται πολύ κοντά με πολύ στενές διαχωριστικές γραμμές. Αν θέλει κανείς να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση, πείτε μα σα παρακαλώ Πώ θέλετε να παρακολύσετε μη συνοδευόμενα παιδιά ανήλικοι, δηλαδή παιδάκια να μπορέσουν αυτό το πύχη σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση να τον ξεπεράσουν και να μπουν στην Ευρώπη. Πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο και θα προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά δίνοντας την δυνατότητα να έρθουν στην Ευρώπη. Είπατε ότι πρέπει ο κίνδυνος λέει να μειωθεί για αυτά τα παιδιά. Πώς θα το καταφέρετε αυτό, πώς θα το πετύχετε. Πραγματικά ενηγματώδες για μένα, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Τρίτο σημείο, πάντα ήμουν υπέρ μιας κοινή πολιτικής για το άσυλο στην Ευρώπη. Θετικό το έβρισκα πάντα αυτό. Πρέπει να εναρμονιστούν τα πράγματα. Αλλά να μιλήσουμε για προδιαγραφές τότε παρακαλώ. Ανησυχώ πάρα πολύ τι θα γίνει σε σχέση με τον ρόλο του προγράμματος ε, της Στοκχόλμης και ποιο ρόλο θα διαδραματίζει η σύμβαση της Γενέβης. Πώς από τη μια μεριά Frontex, ενίσχυση εσωτερικής λέει και εξωτερικής ασφάλειας, όλα αυτά και από την άλλη πλευρά να λέτε ναι θέλουμε μια κοινή πολιτική ασύλου στην Ευρώπη να διασφαλιστεί και πώς θα εγγυηθείτε ότι οι πρόσφυγες, οι πραγματικοί πρόσφυγες θα έχουν τα δικαιώματα που θα τους διασφαλίζουν δικαίωμα για άσυλο. Είναι ενηγματώδη όλα αυτά και γι' αυτό πιστεύω ότι η Στοχόλμη ξεπερνά τις παρακάμπτει τη πραγματικότητα και τις ανάγκες μας. Ευχαριστώ. Παπαδοπούλου παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι το πρόγραμμα τη Στοχόλμη είναι πολύ φιλοδόξο. Εσεί, οι κάτοικοι τη Σουηδία πρέπει να είστε πολύ ευτυχεί. και η χώρα σα είναι μια ευτυχισμένη χώρα. Γιατί λόγω τη γεωγραφική τη θέση ζει σε ένα χώρο πραγματικής ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Προέρχομαι κι εγώ από την Κύπρο και όπως έχει πει ο Μαλτέζος και ο Ισπανός και ο Κύπριος συναδελφός μου, τα πράγματα δεν είναι τα ίδια στη Μεσόγειο. Η Μάλτα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η χώρα μου η Κύπρος βιώνουν μεταναστευτικά ρεύματα και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Και εδώ θα πρέπει να εκδηλωθεί η κοινοτική αλληλεγγύη. Δεν την έχουμε δει μέχρι σήμερα. Μιλώντας για την Κύπρο, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Για 35 ολόκληρα χρόνια καταπατούνται στο νησί μου ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνεται ένας παράνομος επικισμός. Έρχονται τάχατες οικονομικοί μετανάστες από την Τουρκία και επικίζουν τα κατεχόμενα ευρωπαϊκά εδάφη της χώρας μου. Διερωτούμε σε αυτήν την περίπτωση πώς εκδηλώνεται η κοινοτική αλληλεγγύη στο Αιγαίο υπάρχουν παρενοχλήσεις των ελικοπτέρων της Frontex από τουρκικά ε, αεροπλάνα. Διερωτούμε πώς εκδηλώνεται εκεί η κοινωτική αλληλεγγύη. Και το ερώτημα μου είναι το εξή. Για 35 ολόκληρα χρόνια στη χώρα μου υπάρχει καταπάτηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ προσωπικά είμαι πρόσφυγας από την κατεχόμενη περιοχή και δεν μπορώ να επισκεφτώ το σπίτι μου αν δεν επιδείξω διαβατήριο όταν μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη, δείχνοντα μόνο την ευρωπαϊκή μου ταυτότητα. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, πώ εκδηλώνεται η κοινοτική αλληλεγγύη και τι προτίθεται να πράξει η Σουηδική Προεδρία, ώστε να μην μείνουμε μόνο σε διακηρύξει, αλλά έμπραχτα όσοι παραβιάζουν ευρωπαϊκές αρχές να τιμωρούνται. Η Τουρκία πρέπει να λογοδοτήσει γιατί ανέχεστε να κάνει τώρα τη συμφωνία διαπραγματεύση για να επιστρέφουν στην Τουρκία οι λαθρομετανάστε, λίγε μέρε προτού κρυθεί η Τουρκία το Δεκέμβριο του 2009 και δεν έγινε αυτό από το 2002. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύντομα πριν από τα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τις επεξηγήσεις. Φυσικά υπάρχει εδώ λόγος για τον οποίο αυτή η συνεργασία ε, που επιθυμούμε να διασφαλιστεί. Υπάρχουν λόγοι, έχουμε όμως διαφορετικές απόψεις σίγουρα όταν έρχεται η ώρα για δικαιώματα και τον προσδιορισμό έκφραση αλληλεγγύης. Συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και αυτό δημιουργεί και θα δημιουργεί προβλήματα. Κατά τα άλλα θα ήθελα το ερώτημα της κυρίας Ιντφέλτ για τα προσωπικά δεδομένα και την αποθήκευσή τους ε, να ανέφερα, αλλά θα μπορούσα να αναφέρω κάτι διαφορετικό. Είναι ένα σημείο το οποίο με ενδιαφέρει και με αφορά άμεσα και που και για την ίδια τη Σουηδία είναι σημαντικό η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών είναι κάτι σημαντικό και προβλέπει ότι η ευημερία των παιδιών θα πρέπει πάντα να είναι πρώτη ως προτεραιότητα. Διαρωτώ με και με κάπως σε σχέση με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ότι δεν προσδιορίζονται σαφέστερα τα δικαιώματα των παιδιών. Ναι, λέγεται κάτι για τα δικαιώματα των παιδιών, για τα παιδιά, αλλά όχι τόσο εξειδικευμένα και ρητά και κατηγορηματικά. Πρέπει αυτό να είναι σαφέστερο. Ο κύριος Μπόντς παρακαλώ τελευταίο. Eh, Σας ευχαριστώ επιτρέψτε μου να πω ότι Ευχαριστώ για την παρουσίαση και την παρουσία των Σουηδών από πλευρά ε, τη Προεδρία. Πρέπει να πω ότι όταν είχε γίνει παρουσίαση από πλευρά Υπουργού είχα ανησυχήσει. Τώρα ανησυχώ ακόμα περισσότερο. Να σα εξηγήσω γιατί. Η μαζική μετανάστευση κατά τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε μια καταστροφή, σε μια ολέθρια κατάσταση ε, σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη. Δείτε τι γίνεται στην Σουηδία. Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τι πόλει. Το ίδιο ζούμε και στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι ε, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες ε, εγκαταλείπουν οι κάτοικοι του κέντρου ε, λόγω μετανάστευσης τα, τις, ε, ε, τα σπίτια τους. Μπορώ να σας πω ότι μια σημαντική Ολλανδική εφημερίδα πριν από κάποιες εβδομάδες εξέτασε το θέμα αυτό και καταδείχθηκε ότι μαζική μετανάστευση στην Ολλανδία κόστησε δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν λέτε όμως ότι είναι καλή μετανάστευση για την κρίση της οικονομίας μας, αυτό δεν αληθεύει και δεν είναι καλό και δεν ευσταθεί διότι έχουμε πρόβλημα, δημιουργείται τεράστιο κόστος και δεν αποβαίνει υπέρ των ανέργων. Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Η μαζική, η μαζική μετανάστευση δεν αντιμετωπίζει την υπεργύρανση του πληθυσμού μας, διότι και οι μετανάστες αυτοί κάποτε θα γεράσουν, αυτοί που θα έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. στην ε, Ολλανδία ή στη Σουηδία πόσους κατοίκους πρέπει να έχουμε, Εκατό εκατομμύρια κατοίκους για να αντιμετωπίσουμε την υπεργύρανση. Σταματήστε πια τη μετανάστευση, φτάνει πια πρέπει να πω. Ε, Ακούσαμε τις ερωτήσεις αυτές, ε, οι οποίες ε, ήταν ιδιαίτερα ε, ζωντανές. Έγινε ένας πολύ καλός διάλογος και πραγματικά δείχνει η σειρά αυτή ερωτήσεων πόσο πολύ ενδιαφέρονται οι βουλευτές για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Θα ακούσουμε τις απαντήσεις καταρχάς από τον κύριο Γκράνερ και συνέχεια από την κυρία Λούγκρεν. Κύριε Γκράνερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά και θα προσπαθήσω να απαντήσω τις περισσότερες ερωτήσεις η Σουηδία είναι μια μικρή χώρα στα περιθώρια κάπως της Ευρώπης, αρκετά μακριά όπως κάποιος είπε και νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον το να ακούσει κανείς η συζήτηση αυτή γιατί αντικατοπτρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο η πολιτική συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στην Ευρώπη αντικατοπτρίζεται επίσης πάρα πολύ καλά η συζήτηση που γίνεται σε όλα τα πολιτικά κόμματα, σε όλες τις χώρες και εκφράστηκαν όλες οι διαφορετικές πολιτικές απόψεις που εκφράζονται και από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να δώσω κάποια παραδείγματα γιατί προφανώς δεν γίνεται να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ορισμένοι βουλευτές αναφέρθηκαν στην προστασία των δικαιωμάτων και ορισμένοι βουλευτές ζήτησαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία. Και τα δύο αυτά σημεία, ζητήματα, είναι σωστά. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μία ισορροπία. Στην όλη αυτή εξίσωση ποια είναι η θέση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα πράγματα δεν είναι πολύπλοκα για μένα. Υφίστανται τα θεμελιώδη δικαιώματα, ισχύουν για όλους τα κληρονομούμε τα δικαιώματα αυτά, μας τα δίνει ο Θεός, η φύση, οτιδήποτε θέλετε να πιστεύετε, πάντως υφίστανται τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ορισμένα από αυτά δεν είναι καν σχετικά, λένε απόλυτα, κάποια όμως μπορεί να σχετικοποιηθούν κιόλας. Για παράδειγμα, έχω το δικαίωμα να κυκλοφορώ ελεύθερα στους δρόμους. Αν όμω διαπράξω ένα έγκλημα, θα με κλείσουν στη φυλακή και το δικαίωμά μου να κυκλοφορώ ελεύθερα στον δρόμο θα περιοριστεί, έτσι δεν είναι. Μπορώ, έχω να ξεκινήσω, μπορεί να αρχίσω να προγραμματίζω μια τρομοκρατική πράξη. Αν αρχίσω, να, αρχίσω να κάνω κάτι τέτοιο, τότε το κράτος έχει κάθε δικαίωμα να με σταματήσει, να με εμποδίσει. Ορισμένα δικαιώματα λοιπόν είναι απόλυτα, άλλα δικαιώματα είναι σχετικά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να πετύχουμε την απαραίτητη ισορροπία. Ορισμένοι βουλευτέ από ό,τι φάνηκε θέλουν μεγαλύτερη αστυνομική συνεργασία, άλλοι πάλι βουλευτέ ζητάνε μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτή είναι ακριβώ η πρόκληση που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τόσο εσεί στην Επιτροπή σα όσο και εμεί στο Συμβούλιο. Α είμαι τώρα συγκεκριμένο για κάποια ζητήματα. Όσον αφορά την κατάσταση στη Λετωνία, είναι σαφές εδώ ότι όλα τα κράτη-μέλη καλούνται να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα που περιέχονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Ορισμένοι βουλευτές ζήτησαν ένα πιο στεναρό κείμενο για την προστασία των παιδιών, των γυναικών. Συμφωνώ μαζί σας. Θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο για τις ευάλωτες αυτές ομάδες. Θα μπορούσα να αφαιρθώ σε πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση, τα επιχειρήματα, οι ερωτήσεις μιλούν από μόνες τους. Κατέγραψα όλα αυτά τα οποία είπατε εδώ στην Επιτροπή σας και θεωρώ ότι βρίσκεστε πραγματικά στο κέντρο της συζήτησης. Έτσι ακριβώς διαμορφώνεται και η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκράνερ. Το λόγο τώρα έχει η Υφυπουργός Πολιτικής Ασύλου και Μετανάστευση κυρία Λούγκρεν θα γνωρίζετε ότι τέθησαν πάρα πολλά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε ξεχωριστά σε κάθε ερώτημα. Προσπαθήστε δυνατόν να δώσετε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες στη συζήτηση που ήδη έχει λάβει η χώρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι ένα ζήτημα, ένα θέμα που αναφέρθηκε από τις, τους περισσότερους στις παρεμβάσεις τους ήταν το θέμα της αλληλεγγύης. Αυτό το στοιχείο, η αλληλεγγύη, στις συζητήσεις που κάναμε το Σεπτέμβριο από τα κράτη-μέλη επανειλημμένα διαρκώς αναφερόταν το θέμα της αλληλεγγύης. Και όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Γκράνερ, είμαστε φυσικά μια μικρή χώρα, μικρότερη χώρα τη Βόρεια Ευρώπη. Όμως έχουμε και την δική μας πείρα όσον αφορά θέματα μετανάστευσης. Το 2007 είχαμε 37.000 ετούντες άσυλο. Και αν όλα αυτά τα θέσει κανείς σε αναλογία και τα δει αναλογικά, στην Ιταλία 250.000 ετούντες άσυλο θα σήμαινε αυτό σε σχέση για παράδειγμα με τον αριθμό κατοίκων της Ιταλίας εφόσον η αναλογία ήταν από τον αριθμό κατοίκων της Σουηδίας για μας. Και θέλω να υπογραμμίσω με αυτό ότι για μας τα προβλήματα της Μεσογείου, του χώρου της Μεσογείου είναι κάτι που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα. Πολλοί τα προανέφεραν, το προανέφεραν αυτό. Ο Τομπίας Μπίτστρομ, ο υπουργό για θέματα μετανάστευσης, ο ίδιος, τον Ιούνιο είχε πάει στη Μάλτα προσωπικά και είδε τι συμβαίνει εκεί ο ίδιος, η δυσόμαση. Και γνωρίζουμε λοιπόν τα προβλήματα επιτόπου. Όμως οι λύσεις δεν είναι απλές και η επίλυση των προβλημάτων δεν είναι απλή υπόθεση. Η συζήτηση απόψε εδώ το κατέδειξε. Απλές λύσεις, γοριέ, ταχύτατες λύσεις δεν υπάρχουν. Αν κάποιο έχει κάποιο τέτοιο, κάποια τέτοια μαγική συνταγή, να μα την πει, είμαστε ευγνώμονε, να την ακούσουμε. Χρειαζόμαστε κατά τα άλλα όμω μια ισορροπημένη πολιτική. Χρειαζόμαστε βράχη πρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα στη φύση του ένα βραχυπρόθεσμο όσον αφορά το χαρακτήρα του στοιχείο οδηγεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δράσουν το πιλωτικό ακριβώς πρόγραμμα στην Μάλτα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα, απόρρια των συμπερασμάτων της συνάντησης του Ιουλίου. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω και κάτι άλλο. Με τον πιο διαφορετικό τρόπο μπορεί κανείς να εκφράσει και να δείξει την αλληλεγγύη του. Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα, υπάρχουν το Ταμείο Προσφύγων για παράδειγμα, ε, το Ταμείο για τη Συνοριακή Δράση, το Ταμείο για την Υποστήριξη της Παλινόστησης, της Επιστροφής. Ε, ε, τέτοιου είδους μέσα έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα με άλλες συνιστώσεις σε σχέση με πάλι με την συνάντηση κορυφής του Ιουλίου που είχαμε. Οι συναντήσεις δηλαδή οι σχέσεις σε σχέση με τα κράτη προέλευσης και τα κράτη διέλευσης διαμετακόμισης για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να βελτιωθούν. Με την Τουρκία για παράδειγμα, με τις χώρες προέλευσης αυτών των ανθρώπων. Πολλά γίνονται και ο Επίτροπος Μπίλστρομ κατά τη διάρκεια ε, του φθινοπόρου θα επισκεφθούν τις χώρες αυτές, μεταξύ αυτών και την Τουρκία. Πρέπει να βελτιωθούν λοιπόν οι σχέσεις μας ε, σίγουρα και πρέπει να καταφέρουμε αυτές τις χώρες να τις βοηθήσουμε σε σχέση με την ανάπτυξη του δυναμικού τους και των ικανοτήτων τους. Από την άλλη πλευρά, το θεωρώ αποφασιστική σημασία, αν θέλουμε να είμαστε επιτυχεί στη δράση μας, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μακρόχρονα να δράσουμε. Πρέπει αυτή την σφαιρική προσέγγιση να την εντείνουμε πολύ περισσότερο. Πρέπει να υπάρξει διασύνδεση που θα διασφαλίσουμε και θα δράσουμε αποτελεσματικά με τα θεμελιώδη στοιχεία που αφορούν τη μετανάστευση πρέπει να δράσουμε όσον αφορά τις χώρες προέλευσης αυτών των ανθρώπων, των μεταναστών και τις χώρες διέλευσης. Πολλά από αυτά τα μέτρα είναι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα άμεσα μέτρα ώστε να επιληθούν, να αντιμετωπιστούν άμεσα ε, οξύτατα προβλήματα. Για παράδειγμα, στον χώρο της Μεσογείου, για παράδειγμα, Πρέπει όμως να πάμε πιο βαθιά από το επιφανειακό αυτό επίπεδο. Πρέπει μακροπρόθεσμα, σε ένα μακροπρόθεσμο με μακρύτερο χρονικό ορίζοντα ε, πλαίσιο να δράσουμε. Αναφέρθηκε η Frontex πιο πριν και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο σίγουρα. Και από την άλλη πλευρά όταν πρόκειται για το τι μπορεί κανείς να κάνει ώστε απλά να σώσει ανθρώπινες ζωές ε, τότε η Frontex έχει σίγουρα αποφασιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. Στι συζητήσει τον Σεπτέμβριο κατέστη σαφέ επίση ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι η Frontex μπορεί πολλά περισσότερα να πράξει και πρέπει να το ζητήσουμε αυτό, να το καταφέρει. Εδώ όμω τα κράτη-μέλη θα πρέπει τα ίδια να αποφασίζουν τι πόρους, τι κονδύλια, ποιο υλικό και με ποιο τρόπο θα πρικοδοτήσουν και θα ενισχύσουν τη Frontex για να δρά αποτελεσματικότερα. Ένα άλλο στοιχείο. Έχουμε και διαφορετικές απόψεις στη συνέχεια όσον αφορά την οικονομική μετανάστευση. Ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις. Εντάξει. Και αυτές οι διαφορετικές τοποθετήσεις τι δείχνουν. Δείχνουν φυσικά και κάτι άλλο. Δείχνουν πόσο διαφορετικά είναι τα συμφέροντα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη και να καλυφθούν. Το εύρος λοιπόν είναι πολύ μεγάλο των απόψεων και των θεωριών. Μία ενιαία αφετηρία για το σύνολο του προγράμματος της δράσης της Στοκχόλμης είναι για μας ως Σουηδική Προεδρία και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα στοιχείο η καλή αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων μετανάστευσης που πρέπει να αποβαίνει προς όφελος όλων. Δεν, θέλουμε εδώ μόνο τα καλά να επιλέγουμε και να αγνοούμε τις αρνητικές πτυχές, να κάνουμε μια, α ε, ας το πω έτσι, κατεπιλογή αντιμετώπιση θεμάτων. Όχι μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων μετανάστευσης μπορεί να είναι προς όφελος όλων και για τις χώρες προέλευσης αυτών των μεταναστών αλλά και για τις χώρες μετανάστευσης όπως τις δικές μας χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στην Ευρώπη όπως προανέφερα στους μετανάστες αυτούς. Τώρα η Σουηδική Προεδρία ίδια τι κάνει Ελπίζει η Σουηδική Προεδρία ότι η νομοθεσία μας, το νομοθετικό μας έργο για την αγορά εργασίας, για παράδειγμα, το σουηδικό, πρότυπο μπορεί να είναι, το σουηδικό μοντέλο μπορεί να είναι ένα πρότυπο. Έχουμε ένα καλό σύστημα για θέματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και για μετανάστες. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρότυπο. Και εξάλλου έγινε αναφορά και αυτό οι συζητήσεις ε, και πρέπει σίγουρα να εξετάζεται η νομική ασφάλεια, η βεβαιότητα νομικού πλαισίου και νομικών ζητημάτων πρέπει να διασφαλίζεται πάντα. Ταυτόχρονα είναι αυτό ένα σημαντικό εργαλείο, ένα σημαντικό μέσο, ένα σημαντικό στοιχείο στην διαδικασία θεμάτων ασύλου. Μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Διότι αν θέλουμε να έχουμε ένα λειτουργικό κοινό σύστημα για θέματα ασύλου στην Ευρώπη, τότε πρέπει από την άλλη πλευρά να διασφαλίζουμε ότι εκείνοι οι οποίοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να διαμένουν στην Ευρώπη θα πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες τους. Αυτό είναι αυτονόητο και πρέπει να διασφαλίζεται. Πρέπει όμως με τον σωστό τρόπο νομικά να εξετάζεται και να εκτελείται σε ένα νόμιμο πλαίσιο. Τώρα, για τα παιδιά, για τα δικαιώματα των παιδιών ένα πολύ ακαθόδες ζήτημα και δυσχερέστατο θέμα. Γνωρίζετε ότι και στην Υπουργική Συνάντηση πριν από ένα μήνα συζητήθηκε το θέμα θα ε, εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης ε, και θα το υποβάλουμε κατά τις αρχές του 2010. Αναφέρθηκε και το γραφείο η υπηρεσία υποστήριξης ε, για θέματα ασύλου αυτή η υπηρεσία έχει αποφασιστικό ρόλο ώστε στην ε, πρακτική συμφή συνεργασία να μπορέσουμε να προοδεύσουμε, να, κάνουμε, να σημειώσουμε πρόοδο και να μπορέσουμε να ε, συγκροτήσουμε αυτή την υπηρεσία. Απευθύνω έκκληση προς όλους να συνεχίσουμε τη δουλειά μας προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτόν τον στόχο. Η κοινή υπηρεσία υποστήριξη ασύλου είναι αποφασιστική σημασία. Λοιπόν, όπως σας προείπα, υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Αυτές νομίζω ήταν οι σημαντικότερες από αυτές που εξέθεσα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο υπουργού για τις παρουσιάσεις τους, για τις απαντήσεις που δώσανε, στις ερωτήσεις που θέσατε. Καταλήγοντας, θα ήθελα να σε επενθυμίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού μας, του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μία κοινή έκθεση έχει αποσταλεί από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, την Επιτροπή ΑΦΚΟ και την Επιτροπή Ιούρι, δηλαδή νομικών θεμάτων και σταγματικών υποθέσεων, όσον αφορά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ακόμα λοιπόν έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας και βασιζόμαστε σε εσά και για λόγους διαφάνειας θα θέλαμε και περισσότερες πληροφορίες από τη Σουηδική Προεδρία σε σχέση με τη σημερινή συζήτηση Θέλουμε λεπτομερείς απαντήσεις σε κάθε ερώτηση που υποβλήθηκε, γιατί σίγουρα αυτό θα μας βοηθήσει στο να κάνουμε καλά και έγκαιρα τη δουλειά μας. Προβλέπεται για τις 12 Νοεμβρίου ε, να γίνει ψηφοφορία ε, για το πρόγραμμα της Στοκόλμης εδώ στην Επιτροπή μας και στη συνέχεια αργότερα τον Νοέμβριο θα ψηφιστεί το πρόγραμμα αυτό και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας καλώ λοιπόν να μας στείλετε τις περαιτέρω αυτές πληροφορίες και απαντήσεις και όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε εμείς για την κατάρτιση της δικής μας έκθεσης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μας επιτρέψετε να επιτελέσουμε σωστά και εγκαίρως τη δική μας δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ πολύ για να προχωρήσουμε και στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Σημείο 28 με θέμα το δικαίωμα σε διερμηνία και μετάφραση κατά τις ποινικέ δίκες. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ καθίστε. Έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας. Καθείς, παρακαλώ πολύ. Η κυρία Ντβέλ θα αναλάβει την Προεδρία γιατί έχω κάποιες άλλες συνειδημένες υποχρεώσεις που πρέπει να αποχωρήσω. Η κυρία Ντβέλ λοιπόν θα προεδρεύσει για το υπόλοιπο της συνεδρίασης και θα καλύψει το ζήτημα 28 δικαίωμα στη και μετάφραση κατά τις ποινικές δίκες. Great. If I cannot, the floor is all yours. Thank you very much. I think the next point on the agenda is the report of Sarah Ludford on the right to interpretation. Θα μιλήσουμε τώρα για το δικαίωμα σε διερμηνία και μετάφραση κατά τις ποινικές δίκες. Θα πρέπει να διαβάσω μια σύντομη ε, εισαγωγή μου, είπανε πρωτού δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και αρκετό καιρό επιθυμεί να εγκριθεί ένα νομικό μέσο για τα δικαιώματα του εναγωμένου. Μια πρώτη απόπειρα έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν λειτουργήσε γιατί τα κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε σχέση με μια πρόταση απόφαση πλαισίου που, προτάθηκε το 2004. Γίνονται τώρα διαπραγματεύσει για μια δεύτερη πρόταση απόφαση πλαισίου, όπου θα ακολουθηθεί μια προσέγγιση βαθμιαία, βήμα προ βήμα, και το πεδίο εφαρμογή εδώ πέρα είναι πιο περιορισμένο. Αναφερόμαστε μόνο στο δικαίωμα δερμηνία και μετάφραση. Επίση, η Σουηδική Προεδρία, που θεωρεί ότι τα δικαιώματα του αγωμένου είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα πρότεινε κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου τα οποία θα συνοδεύουν την έγκριση της απόφασης πλαισίου και έχει ξεκινήσει επίσης και την επεξεργασία ενός οδικού χάρτη για την ενίσχυση των δικαιωμάτων αγωμένου στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών. Θα ήθελα να δώσω καταρχώς το λόγο στη Βαρόνη Σάρα Λάτφορντ και συνέχεια σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προεδρίας. Σάρα Λάτφορντ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εν μέρη κάνετε ένα μέρο τη δική μου τη μέσω τη εισαγωγή σα αυτή. Πρέπει να σας πω βέβαια τα πράγματα είναι κάπως χειρότερα από ό,τι τα παρουσιάσατε. Πριν από 10 χρόνια ξεκίνησε όλη η προσπάθεια να έχουμε τουλάχιστον μία πρόταση για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του εναγωμένου. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια τον Ιούλιο του 2000 μέσω ανακοίνωσή τη για την αμοιβαία αναγνώριση των τελικών αποφάσεων σε ποινικέ υποθέσει, είπε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η μεταχείριση των υπόπτων αλλά και, δηλαδή ο ενάγων και ο ενασγόμενος δεν θα πρέπει να πλήττονται στα πλαίσια της αμοιβαία αναγνώρισης και ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερες διασφαλίσεις στα πλαίσια της ποινική διαδικασίας. Αυτή λοιπόν ήταν η αρχική απόπειρα που είχε γίνει και στη συνέχεια ακολούθησαν διάφορα μέτρα τα οποία λέγαν ότι η αμοιβαία αναγνώριση εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους που ουσιαστικά καθορίζουν την αποτελεσματικότητά της και ένας, μία από αυτές τις παραμέτρους είναι η εξασφάλιση των δικαιωμάτων και των υπόπτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή έδειξε τον δέοντα ενθουσιασμό, υποστήριξε τις προτάσεις αυτές και θέλησε να εγκριθεί ένας τέτοιος μηχανισμός. Είδαμε διάφορα μέτρα τα οποία ενισχύουν την διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία και τη συνεργασία των εισαγγελικών αρχών αλλά μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι αρκετά ανισόρροπα θα έλεγα, γιατί από τη μια έχουμε τα μέτρα αυτά, αλλά δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα αμοιβαία εμπιστοσύνη όσον αφορά τον εναγόμενο. Ουσιαστικά προασπίζουμε μέχρι στιγμής περισσότερο τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Το 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα μετά από πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνέχεια το 2005 με την ε, έκθεση Buchenwald. Θα γνωρίζετε η παλαιότερη εδώ πέρα όλη αυτή τη διαδικασία. Είχε τοποθετηθεί πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχε προταθεί και τότε μία απόφαση πλαίσιο την άνοιξη του 2004 συγκεκριμένα. Είχαμε ολοκληρωμένη τότε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου προβλεπόταν μία δέσμη μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των αγωμένων. Ακόμα και στην έκθεσή μας τότε, στο ψήφισμά μας τότε, είχαμε πει ότι η προτενόμενη απόφαση πλαίσιο αποτελούσε ένα, ένα πρώτο μόνο βήμα προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα μειόμορφο σύστημα προάσπισης των δικαιωμάτων των αγωμένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ούτε και τότε είχαμε θεωρήσει ποτέ ότι η πρόταση αυτή από μόνη της αρκούσε. Αυτό που συνέβη όμως τελικά με την πρόταση αυτή είναι ότι βρήκε πολύ στεναρή αντίδραση από το Συμβούλιο το 2007 όταν πολλά μέλη τότε του Συμβουλίου είπανε ότι δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν μια τέτοια πρόταση. και ανάλογη προσπάθεια έγινε και με μια πρόταση ψηφίσματος να δημιουργηθεί δηλαδή μια μη δεσμευτική πρόταση, να υπάρχει τουλάχιστον ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα που να καταχειρώνει τρόπον τεινά τα δικαιώματα αυτά. Πάρα πολλοί ευρωβουλευτέ είχαν τότε παραπονεθεί για τη στάση αυτή του Συμβουλίου και πάρα πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και το κενό αυτό έχει οδηγήσει σε πάρα πολλά προβλήματα βέβαια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πέρυσι άκουσα ότι ένας υψηλά ιστάμενος αστυνομικός στην Αγγλία είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης όχι μόνο για αποδεδειγμένα εγκλήματα αλλά ακόμα και για απλή διερεύνηση, απλή ανάκριση. Και Νομίζω ότι και αυτό το ζήτημα, προβλήματα τα οποία κρεμούν δηλαδή και υπάρχουν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψη, θα πρέπει να επιληθούν. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν δεν προασπίζονται σωστά τα δικαιώματα του εναγωμένου. Δεν προβλέπονται καθόλου τα δικαιώματα του εναγωμένου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Σύλληψης. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να επιθυμούμε να ξαναξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία και να καταφέρουμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των αγωμένων στις ποινικές διαδικασίες. Πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε την Σουηδική Προεδρία γιατί αν μη τι άλλο έχει πολύ καλές προθέσεις. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια πολύ καλή δέσμευση από τη Σουηδική Προεδρία, στα πλαίσια του προγραμματός της δηλαδή, και η βασική ιδέα εδώ πέρα είναι να έχουμε έναν οδικό χάρτη. Όλα ονομάζονται πλέον οδικό χάρτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να κάνουμε και να έχουμε μεμονωμένες ξεχωριστές αποφάσεις πλαίσιο από το να έχουμε μία κοινή όπως προσπαθήσαμε να κάνουμε στο παρελθόν. Και θα υπάρχει και ένα ψήφισμα στο οποίο θα προβλέπεται ακριβώς η πρόθεση αυτή να καταλήξουμε σε πέντε αποφάσεις πλαίσιο και φαντάζομαι μάλλον θα έχουμε και μία πράσινη βίβλο όσον αφορά την κράτηση των υπόπτων δηλαδή. Ο δικός χάρτης θα περιέχει και μία πτυχή που θα έχει να κάνει με τη συνεργασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής δεν έχει προταθεί καμία διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον οδικό αυτό χάρτη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτή η δέσμευση για συνεργασία με το Κοινοβούλιο παραμένει κάπως κενή. Πάντως, θα έχουμε αυτό το σφαιρικό δικό χάρτη, ξεχωριστές αποφάσεις πλαίσιο, για την οποία εγώ θα είμαι η συγγήτρια, δηλαδή για την δερμηνή και τη μετάφραση στις ποινικέ δίκες. Και στη συνέχεια η απόφαση αυτή πλαίσιο θα συνοδεύεται από ένα ψήφισμα το οποίο θα περιέχει πιο λεπτομερείς διατάξεις. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα αυτή τη στιγμή. Από το να έχουμε μία πάγια νομοθεσία όπω το παρελθόν, έχουμε ξεχωριστέ αποφάσεις πλαίσιο, εκ των οποίων οι πρώτε τουλάχιστον θα συνοδεύονται από ένα μη δεσμευτικό κείμενο κατευθυντηρίων γραμμών. δεν καταλήγουμε στην ευκταία τελικά λύση, σε αυτό το Ελντοράδο το οποίο είχαμε οραματιστεί στην αρχή, αλλά μη χειροβέλτιστον τελικά. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε ε, με τις ε, υφιστάμενες συνθήκες. Τώρα εναπόκειται σε εμά να δούμε αν ε, τα πράγματα είναι πιο αισιόδοξα, πιο απεσιόδοξα, πιο θετικά, πιο αρνητικά. Εναπόκειται αυτό στην κρίση του καθενός. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα ζητήματα που διευθετούνται στα πλαίσια της απόφασης πλαισίου, αλλά στην πρώτη απόφαση πλαίσιο, μη τι άλλο, προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι νομοθετικές διατάξεις θα καλύπτουν μόνο το δικαίωμα διερμηνίας και μετάφρασης κατά τις ποινικέ διαδικασίες και κυρίως στα πλαίσια των διασυνοριακών ποινικών δικών, δηλαδή όπου μιλάμε για ένταλμα, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Δεν θα ισχύει δηλαδή το δικαίωμα αυτό σε δερμηνία και μετάφραση, τουλάχιστον η απόφαση πλαίσιο για εσωτερικέ δικαστικέ υποθέσει στα πλαίσια ενό κράτου μέλου. Δεν μπορεί να ισχύει, για παράδειγμα, μόνο στο Βέλγιο, αν η υπόθεση είναι καθαρά βελγική και δεν είναι διασυνοριακή. Να συντομεύεται, λέει η Πρόεδρος. Υπάρχουν λοιπόν πολύ εξατομικευμένα και λεπτομερή ζητήματα τα οποία προκύπτουν σε κάθε απόφαση πλαίσιο που θα εγκριθεί και τα περισσότερα από αυτά θα μπορούσαν να επιληθούν ε, βάσει της διακριτικής αυχαίρειας κάθε κράτους μέλους. Θα πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν τελικά πιστεύει ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση και θα, θα πρέπει όντως να ακολουθήσουμε τελικά αυτό το δρόμο ή μήπως τελικά έχουμε μια καλύτερη εναλλακτική λύση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Επομένως, το ερώτημά σας είναι, είναι το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Η κυρία Αντωνέσκου σας ειναι ειναι το ποτηρι μισοαδιο πρώτη στον κατάλογο μιλητών από το ΕΛΚ. Να σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, δεδομένου του γεγονότος ότι πρόκειται για την πρώτη παρέμβαση σε συζήτηση, θέλω να παρουσιαστώ. Είμαι Ιωάννα Αντωνέσκου. Είμαι κοινοβουλευτική εκπρόσωπο από τη Ρουμανία και είμαι σκιώδη εισηγήτρια επίση για αυτά το θέμα αυτή τη έκθεση. Δικηγόρο είμαι το επάγγελμα. Και αυτό είναι ένας ακόμα λόγος, γιατί τα δικαιώματα του πολίτη, του ατόμου, για μένα προσωπικά αποτελούν προτεραιότητα. Θα ήθελα να χαιρετήσω λοιπόν το γεγονός ότι εδώ η Σουηδική Προεδρία στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε να δρομολογήσει τα, τις πτυχές αυτές του εναγόμενου, των δικαιωμάτων του εναγόμενου σε ποινικέ δίκες. Όπως προανέφερε η κυρία Λάτφοντ, υπήρξε λυπής πρόοδος μέχρι σήμερα. Απουσία πρόοδου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει απουσία ισορροπίας όσον αφορά την πρόοδο, όσον αφορά την γενική αναγνώριση θεμάτων ποινικού χαρακτήρα στην ποινική δικονομία και αυτό την αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης των ε, νομολογιών των δικαστηρίων, των αποφάσεων των δικαστηρίων μπορεί να το διακυβεύσει ως θέμα. Μπορεί, ε, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ελάχιστες προδιαγραφές που θα ισχύουν ώστε να υπάρχει η εμπιστοσύνη στην ομολογία και στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Ένας διερμηνέας ε, δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ δύο ατόμων που δεν κατέχουν την ίδια γλώσσα έτσι λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια γέφυρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τα μέλη της Επιτροπής και έχουμε και την Επιτροπή ανάμεσά μας. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη ώστε να υπάρχει έλεγχος της ασφάλειας και της ορθότητας, της διερμηνίας και της μετάφρασης. Διότι ένα ασφάλμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Πρέπει να υπάρχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για αυτούς τους διερμηνείς και μεταφραστές στον τομέα ακριβώς της της ε, νομικής ορολογίας. Θα ήταν ακόμα και ίσως πιθανόν στην Ευρώπη να δημιουργηθεί ένα μητρό διαθέσιμων μεταφραστών και διερμηνέων που κατέχουν τη νομική ορολογία. Διότι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει δυσκολία να βρεθεί έγκαιρα ένας διερμηνέας που θα καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ευχαριστώ. Okay, thank you Σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος και τελευταίος είναι η κυρία Ρομέρο Λόπες, τελευταία. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι επίσης και η συγγήτρια, ε, ε, για αυτήν την απόφαση ε, πλαίσιο, η οποία όπως είπαμε ε, μας ε, ξανα προτείνει ένα θέμα το οποίο απέτυχε το 2004 και αυτό λόγω ενός ε, μπλοκαρίσματος, μιας τροχοπέδησης που υπήρξε σχετικά. Και αυτό γιατί ε, δεν είχαμε καταφέρει να ορίσουμε ποιοι είναι οι ελάχιστοι κανόνες για τα ε, δικαιώματα ε, των, ε, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μία πρόταση η οποία αναφέρεται μόνο στο θέμα της διερμηνίας και της μετάφρασης και έστω και αν πρόκειται για κάτι το εντελώς ε, κατακαιρματισμένο και αυτή δεν είναι η, μόνη διαδικασία μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε να προδεύουμε σε άλλα θέματα συμπεριλαμβανομένου και της ε, χάρτας ε, των δικαιωμάτων Νομίζω λοιπόν ότι η θετική η πρωτοβουλία δεδομένου ότι Τίνουμε προς ελάχιστους κανόνες. Θέλουμε λοιπόν να ρωτήσουμε την Κομισιόν δεν θεωρεί ότι το κείμενο είναι ιδιαίτερα θολό για όσον αφορά ορισμένα σημεία τα οποία καθορίζουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην διερμηνία και τη μετάφραση όταν μιλάμε ε, για ποινική δίκη θα έπρεπε να ορίσουμε σαφώς ποια είναι τα δικαιώματα και η διαδικασία. Αλλά μιλάμε όμως για τον ορισμό μίας και μόνης διαδικασίας. Δεν προχωράμε ιδιαίτερα. Επίσης θέλουμε να ξέρουμε αν υπάρχει διαβάθμιση του δικαίου διότι εξαφανίστηκε ο χάρτης ο οποίος αναφερόταν πρώτα σε αυτό το θέμα. Και όποιος δικάζεται θα έπρεπε να είχε την αναγνώριση αυτής της ε, χάρτας ε, δικαίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος θα ήθελε να παρέμβει Παρακαλώ, όχι. Τότε καλό πρώτα την Προεδρία του Συμβουλίου και μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα να παρέμβουν. <clears throat> Με αυτή τη σειρά κατανόησα ότι θέλετε να παρέμβετε. Εξ ονόματο τη Σουηδική προεδρία, δύο ονόματα έχω εδώ. Ποιο θα παρέμβει. Η κυρία Όμαν, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σα ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Είναι μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση για μένα που βρίσκομαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίδεται ευκαιρία να παρουσιάσω τα σχέδια της Ιδικής Προεδρίας όσον αφορά τα δικαιώματα του ναγωμένου και να σας ενημερώσω για το πώς έχουν τα πράγματα. Θα ξεκινήσω πηγαίνοντας το 2007, τον Ιούνιο του 2007. Την εποχή εκείνη είχαμε ήδη διανύσει τρία χρόνια συζητώντας μία πρόταση για μία απόφαση πλαίσιο όσον αφορά τα δικαιώματα του ναγωμένου. Και η πρόταση αυτή υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2004 και το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2007 έπρεπε να αναγνωρίσει τελικά ότι δεν ήταν δυνατό να καταλήξει σε μια συμφωνία μόλον ότι είχαν περάσει τρία ολόκληρα χρόνια διαπραγματεύσεων, μόλον ότι η Γερμανική Προεδρία και άλλες είχαν υποβάλει πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες. Είχαμε φτάσει σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Έτσι λοιπόν μπήκε σε ένα σιρτάρι η πρόταση αυτή και δεν συζητήθηκε από τότε. Και λίγο καιρό μετά αρχίσαμε να προετοιμάζουμε εμεί τη Σουηδική Προεδρία και γνωρίζαμε ήδη από την αρχή ότι το ζήτημα αυτό θα αποτελούσε προτεραιότητα για τους ειδική Προεδρία. Ιδίω η Μπεατρή Άσκ, η δική μα Υπουργό Δικαιοσύνη που έχει έρθει και στην Επιτροπή σα και σα έχει μιλήσει, είχε πει ότι το ζήτημα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και το ερώτημα που τέθη τότε ήταν πώ μπορούμε εμεί ω ειδική Προεδρία να ξεκινήσουμε πάλι τη συζήτηση για τα δικαιώματα αναγωμένου. Αυτή τη στιγμή όλε οι παρελθούσε προσπάθειε είχαν αποτύχει. Ορισμένα πράγματα ήταν εξ αρχή ξεκάθαρα για μα. Πρώτον, τα δικαιώματα του ναγωμένου είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο για τα κράτη-μέλη. Επομένω, ξέραμε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο το έργο μα. Και δεύτερον, γνωρίζαμε ότι δεν είχαμε δικαίωμα να αποτύχουμε πάλι. Δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε δεύτερη αποτυχία. Και ήταν λοιπόν ξεκάθαρο για μας ότι δεν μπορούσαμε απλώς να ξεσκονίσουμε την παλιά αυτή έκθεση και να την επαναφέρουμε χρειαζόμασταν μία νέα στρατηγική, εντελώς διαφορετική και πιστεύαμε και ακόμα πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε, μάλλον ο μόνος τρόπος για να σημειώσουμε πρόοδο, είναι να αντιμετωπίσουμε τα δικαιώματα εναγωμένου βαθμιαία, βήμα προς βήμα, όπου κάθε φορά θα επικεντρωνόμαστε σε έναν μικρό, περιορισμένο τομέα και θα προχωρούμε έτσι σιγά σιγά Θεωρούμε ότι η προσέγγιση αυτή είναι ρεαλιστική, είναι ακόλουθα και αρκετά φιλόδοξη. Επικεντρωνόμενοι κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο τομέα, μπορούμε να καλύψουμε πλήρως κάθε δικαίωμα, μπορούμε να επισέλθουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες και επομένως για κάθε δικαίωμα που θέλουμε να διασφαλίσουμε μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Προκειμένου όμως η στρατηγική αυτή να είναι και σταθερή και προκειμένου να είναι τελικά και σφαιρική και να έχει μια συνέπεια, και να συνεχιστεί ουσιαστικά και η εργασία μα χρειαζόμασταν μια γενική καθολική συμφωνία. Γι' αυτό το λόγο αναφερθήκαμε τότε στην οδικό χάρτη. Τι είναι ο οδικός χάρτη, Ο δικό χάρτης είναι μια μακροπρόθεσμη πολιτική συμφωνία για να εργαστούμε στα πλαίσια των δικαιωμάτων αγωμένου. Τι γίνεται? Τα κράτη-μέλη ουσιαστικά λένε ότι ναι, πρέπει να επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινότητα και να διασφαλίσει τα δικαιώματα του αγωμένου. Καλείται κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσει για τα ζητήματα που καλύπτουν στον δικό χάρτη, όπου ουσιαστικά θα καλύπτονται όλα αυτά τα οποία είχαμε στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάποια παραπάνω ακόμα ζητήματα. Και επίση στον δικό χάρτη δεσμεύονται τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με τα ζητήματα αυτά ω ζητήματα προτεραιότητας. Και με χαρά μπορώ να σας πω ότι έχουμε ομόφωνη υποστήριξη για τη στρατηγική αυτή από τα κράτη-μέλη. Συνεπώς, την 1η Ιουλίου η Ειδική Προεδρία παρουσίασε τον οδικό αυτό χάρτη. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση απόφασης πλαισίου για το πρώτο ζήτημα, για τη δερμηνία και τη μετάφραση κατά τις ποινικέ δίκες. για τα άτομα επίσης που εμπλέκονται σε υποθέσεις ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Και μερικές μέρες αργότερα η Σουηδική Προεδρία παρουσίασε ένα ψήφισμα όσον αφορά το ζήτημα του δικαιώματος σε δερμηνία και μετάφραση στις ποινικέ δίκες, όπου εμπεριέχονται στο ψήφισμα αυτό πρακτικές διατάξεις για να εφαρμοστεί η απόφαση πλαίσιο. Έτσι λοιπόν αυτή η πρώτη απόφαση πλαίσιο συνοδευόμενη από το ψήφισμα αποτελεί το πρώτο βήμα εφαρμογής του οδικού αυτού χάρτη που θα διασφαλίσει τα δικαιώματα του αγωμένου. Και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να πετύχουμε προστιθέμενη αξία στο ζήτημα αυτό. καταφέρνουμε να καλύψουμε συγκεκριμένα ζητήματα στην απόφαση πλαίσιο και ό,τι δεν μπορεί να περάσει στην απόφαση πλαίσιο μπορεί να βρει τη θέση του ουσιαστικά στο ψήφισμα που θα συνοδεύει την απόφαση πλαίσιο. Βρισκόμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης των τριών αυτών πρώτων κειμένων τελείωσαν οι συζητήσεις στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, έχουν περάσει συζητήσεις σε ανώτερο πλέον πολιτικό επίπεδο και θέλω να σας πω ότι τα πράγματα προχώρησαν πολύ γρηγορότερα από ό,τι τολμούσαμε ποτέ να φανταστούμε στην αρχή της διαδικασίας. Οι συζητήσεις ήταν απόλυτα επικοδομητικές και τα κράτη-μέλη επιθυμούν όντω να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, σε θετικά αποτελέσματα αυτή τη φορά. Έχουμε διανύσει λοιπόν πολύ σημαντικό δρόμο από το 2007. Συμβουλευτήκαμε επίση και το Συμβούλιο τη Ευρώπη, το οποίο γνωμοδότησε και για τον οδικό χάρτη και για την απόφαση πλαίσιο και για το συνοδευτικό ψήφισμα και φροντίσαμε να λάβουμε υπόψη πολλέ από τι παρατηρήσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη, οι συζητήσει που γίνανε στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Φιλοδοξία μας και στόχος μας είναι να εγκριθεί, επεμβαίνει πρόεδρος, μπορείτε σιγά σιγά να καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα. Ναι, ναι, αυτό κάνω τώρα, λέει η ομιλήτρια. Στόχος μας και φιλοδοξία μας λοιπόν είναι να εγκριθεί στις 23 Οκτωβρίου δικός χάρτη και στη συνέχεια τόσο απόφαση πλαίσιο όσο και η συνοδευτική ψηφοφορία, το πρώτο δηλαδή βήμα της διαδικασίας, να εγκριθεί από πολιτικής πλευρά την ίδια ημέρα και στη συνέχεια θα περάσουμε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προσλέπω ιδιαίτερα στη συζήτηση που θα γίνει και στη γνωμοδότηση που θα υποβάλλετε. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστώ. Πρωτού δώσω τον λόγο στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποια λεπτά. Μπορώ να σας ρωτήσω, κατανοήσαμε σωστά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ζητήθηκε να διαβουλευτεί επ' αυτού του οδικού χάρτη, ενώ ζητήσατε να διαβουλευτεί το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σωστά το κατανόησα. Ναι, διαβουλευτήκαμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά έχουμε υποβάλει και το, την απόφαση αυτή για διαβούλευση και στην Ευρωβουλή σύμφωνα με τους κανονισμούς της συνθήκης, με τα όσα προβλέπονται από τη συνθήκη. Αληθεύει. Λοιπόν και πάλι, διαβουλευθήκατε για τον οδικό χάρτη το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απόφαση πλαίσιο. Αληθεύει αυτό, σωστό. Ναι, σωστό. Εντάξει, ευχαριστώ. ήθελα να αποσαφινιστεί αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα τώρα παρακαλώ. Διότι έχω τον μη επίζηλο ρόλο τον αντιπαθητικό ρόλο να είμαι αυστηρή και να διασφαλίσω ότι θα τελειώσουμε έγκαιρα. Να είστε σύντομοι λοιπόν παρακαλώ, το επαναλαμβάνω. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε για την παρουσίαση αυτή. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ την ε, Βαρονέσα. Εσείς και η Προεδρία κάλυψαν ούτως ή άλλως, ε, καλύψατε αυτά τα οποία θα ήθελα να πω και έτσι σε σχέση με την απάντηση κάποιων πραγμάτων, δύο λόγια θα ήθελα να πω πρώτα εισαγωγικά. Προσωπικά με ικανοποιεί ιδιαίτερα να είμαι στην, στην ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ παρουσιάζοντας αυτά τα θέματα των δικαιωμάτων των εναγωμένων. Τα τελευταία χρόνια είχα εμπλακεί έντονα σε αυτό το έργο και η πρώτη φορά που προσήθα να προσφωνήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν το 2003 όταν παρουσιάσαμε την, την πράσινη βίβλο από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Δικαιώματα Εναγωμένων. Και σε αυτή τη διαβούλευση καταδείχθηκε ότι υπήρχε υψηλότατο βαθμό υποστήριξη για αυτό το έργο. Αυτό ο βαθμό υποστήριξη δεν μειώθηκε ποτέ, δεν υποβαθμίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τα διάφορα κράτη-μέλη, από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει κτλ. Είμαστε λοιπόν δεσμευμένοι για ελάχιστε κοινέ προδιαγραφέ. Και εμεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι είναι απόλυτη σημασία, πρωταρχική σημασία αυτό για να μπορέσουν τα πράγματα να λειτουργήσουν σωστά. Και αυτό επαληθεύτηκε και επιβεβαιώθηκε σε μια μείζωνα μελέτη που συντάχθηκε από το ε, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, ε, ULB, Université Libre de Bruxelles. Όλοι όσοι εργάστηκαν στο, εργάζονται στον τομέα του ε, ποινικού δικαίου ομόφωνα συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχουν δικαιώματα και μέτρα που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εναγωμένων. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη φορά να το καταφέρουμε, να πετύχουμε το εγχείρημά μας. Την τελευταία φορά είχε υποβληθεί μια δέσμη δικαιωμάτων για τους εναγόμενους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιστάθηκαν κάποια κράτη-μέλη, υπήρξαν διαφωνίες και έτσι ε, είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση επαρκεί και δεν χρειάζεται αυτή η δέσμη. Είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, η Ευρωπαϊκή Συνθήκη, χρήσιμη πολυσχηδώς και δει την ομολογία του ΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για να κατανοήσει ότι υπάρχουν πολλές ε, παραβιάσεις αυτής της ε, σύμβασης ακόμα όμως. Αυτό που θέλαμε να πούμε είναι ότι δεν είναι κομμένη και ραμμένη η σύμβαση αυτή για τα θέματα της αμοιβαίας αναγνώρισης και αυτό είναι ένα κενό που θέλουμε να καλύψουμε με αυτή τη δουλειά μας. Υποστηρίζουμε ολόθερμα την ε, σουηδική προσέγγιση. Είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα λειτουργούσε η πρόταση με δέσμη μέτρων. Έπρεπε να κατακαιρματίσουμε τα δικαιώματα εναγωμένων σε τμήματα ε, τομεακά. Είναι πολύ πιο εύκολο να διαπραγματευτούμε ένα δικαίωμα κάθε φορά, ένα λάξα και είδαμε ότι όταν ε, υπήρχε η δέσμη, οι ε, κράτη-μέλη συμφωνούσαν στη γενική προσέγγιση, αλλά είχαν πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο δικαίωμα και αυτό του οδηγούσε να τροχοπεδίσουν όλη τη δέσμη. Αν κατακαιρματίσουμε, αν το κατατμήσουμε σε τμήματα, σε σκέλη, τότε μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και υπογραμμίζω και αποδέχομαι πλήρω αυτά που είπε η εκπρόσωπο τη Σουηδική Προεδρία για τι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο. Ήταν αυτή τη φορά πολύ πιο επικοδομητικές από ό,τι στο παρελθόν. Μέτρο Α, το πρώτο μέτρο για τον οδικό χάρτη, για τα δικαιώματα μετάφρασης και διερμηνίας. Στόχος είναι να αποσαφινιστούν ακριβώς πότε δημιουργούνται τέτοια δικαιώματα, πότε αυτό το δικαίωμα στοιχειοθετείται. Υπήρχε θέμα για την διατύπωση και θα επανέλθω στο θέμα αυτό και θα τοποθετηθώ επ' αυτής της διατύπωσης τώρα. Είναι σαφής η διατύπωση. Καθορίζει σαφώς και με σαφήνεια πότε υπάρχει δικαίωμα για διερμηνία. Συζητούμε κάποια από αυτά τα θέματα αλλά είναι αρκετά, είναι πολύ συγκεκριμένο όταν αφορά δικαιώματα εναγωμένου στη διερμηνία. Και το ίδιο και για τη μετάφραση. Υπάρχει απαρίθμηση, καθορισμό στην πρόταση, ποια τουλάχιστον έγγραφα πρέπει να μεταφράζονται οπωσδήποτε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι αρκετά συγκεκριμένη και όχι γενικόλογη η διατύπωση είναι σαφής και περιεκτική. Για να ολοκληρώσω με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόλις το μέτρο Α υιοθετηθεί και εγκριθεί, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πολιτική συμφωνία κατά τα τέλη Οκτωβρίου, θα ξεκινήσουμε τη δουλειά στο μέτρο Β, το δεύτερο, το δικαίωμα όσον αφορά τα ε, ε, δικαιώματα να γνωρίζει κανείς ε, τι συμβαίνει σε σχέση με την σύμβαση για την κατηγορία, ποια είναι η κατηγορία. Το Γ θα, καλύπτει την νομική υποστήριξη, συνδρομή και συμβουλή. Το Δ θα, θα είναι το δικαίωμα να μπορεί κανείς κανείς να έχει επαφή με το δικηγόρο του για παράδειγμα ως εναγόμενος κατά τη διάρκεια της κράτησης και με τις προξενικές αρχές. Πρόεδρε, βλέπω πω με κοιτάζετε, θα είμαι ταχύτατη. Και το ε θα είναι προστασία των ιδιαίτερα ευπαθών, ευάλωτων ε, κρατουμένων εναγωμένων. Συγχωρείτε. Απαντώ στις ερωτήσεις. Πρώτα, μία παρέμβαση της Βαρονέσας Λάτφορντ για το αν η πρόταση αυτή θα καλύπτει ποινικέ διαδικασίες και ε, ή όχι καλύπτει και ε, ποινικέ ε, διεργασίες ε, και εγχώριες δικαστικές υποθέσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει υψηλό βαθμός συνένεση από τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό, να καλύπτονται αυτές οι δύο πτυχέ. Είμαι ευελπιστώ λοιπόν ότι αυτή τη μορφή θα πάρει η τελική, το τελικό μέσο όταν θα εγκριθεί όταν θα υπάρξει έγκριση. Πώς μπορούμε στη συνέχεια, κυρία Αντωνέσκο, Αντωνέσκου στην ερώτησή της, πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να έχουν δοκιμές ε, τεστ για την επάρκεια των διερμηνέων. Έχουμε μια νέα προσέγγιση αυτή τη φορά. Να έχουμε μια νομοθετική πρόταση συν επιπλέον μια πρόταση ψηφίσματος για δεσμευτικά μέσα για τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτή η πρακτική λειτουργεί συνήθως αρκετά καλά, πραγματικά καλά, διότι το μίσο που είναι δύσκολο να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη και που έχουν κάποιες ενστάσεις ή αντιστάσεις τα κράτη-μέλη να συμπεριληφθούν, με αυτό το ψήφισμα για τις βέλτιστες πρακτικές μπορούν να ενδώσουν τα κράτη-μέλη και να αποδεχθούν και να καταφέρουμε έτσι να έχουμε τη τις βέλτιστες πρακτικές με χρηματοδοτική υποστήριξη και συμβουλές για την ε, εκτέλεση και την εφαρμογή αυτού, αυτού του μέσου το ψήφισμα προβλέπει ε, διατάξεις για την κατάρτιση, επιμόρφωση, ε, εκπαίδευση διερμηνέων και σε αυτό το σημείο επίσης συμπεριλαμβάνει και μια διάταξη για ένα μητρό. Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν τέτοιου είδους μητρώα ε, επαρκών διερμηνέων με επάρκεια και αυτό φυσικά μεταξύ των κρατών μελών όπου υπάρχει κοινή γλώσσα, γλώσσα υπάρχει ενθάρρυνση να προαχθεί. Θα είναι ένα νέο μέσο τεχνολογικό το οποίο θα είναι στη διάθεση ακριβώς των αρχών των κρατών μελών ώστε να μπορούν να υπάρχουν ανταλλαγέ αυτών των στοιχείων των μητρών με τον καλύτερο τρόπο. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο της πρότασης ψηφίσματος. Νομίζω απάντησα όλες τις ερωτήσει και προς το συμφέρον της συντομίας ολοκληρώνω εδώ και σταματώ. Σας ευχαριστώ. Thank ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που απαντήσατε τις ερωτήσεις. Και τώρα θα θέλατε να επανέλθετε uh, Σας ευχαριστώ πολύ για τις uh, διασφαλίσεις που μας δώσατε. Να ευχαριστήσω και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζομαι και νέα γυαλιά γιατί διαβάσα καλά το άρθρο 1 για το πεδίο εφαρμογή και με καθυσίχασε το ότι καλύπτονται όλες οι ποινικέ διαδικασίες και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την διόρθωσή σας αυτή. Πιστεύω όμως ότι υφίστανται ακόμα προβλήματα με αυτή τη βαθμία βήμα προς βήμα προσέγγιση. Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να εξετάσουμε σφαιρικά την πρόταση αυτή, ιδίως ε, τις πτυχές που θα έχουν να κάνουν με τη νομική αρρωγή Πώς θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν τελικά όλοι πρόσβαση στο δικαίωμα δερμηνίας και μετάφρασης και πώς θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε και τις ευάλωτες ομάδες. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρετε να καλύψει ομάδες αυτές αν δεν προβλέπετε συγκεκριμένο μέτρο για τις ευάλωτες ομάδες. Όσον αφορά τώρα τον οδικό χάρτη. Ήταν καλό, πολύ καλό κυρία Πρόεδρε, ότι καταφέραμε να διευκρινίσουμε από τη Σουηδική Προεδρία ότι ε, θα μπορούμε να συμμετέχουμε και εμείς στην κατάρτιση του δικού αυτού χάρτη και ότι δεν θα περιοριστούμε σε μία απλή διαβούλευση. Θέλουμε σίγουρα εμείς να έχουμε κάποια αντίγραφα της γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, να δούμε πώς αυτοί συμβούλευσαν το Συμβούλιο για τα ζητήματα αυτά. Ορισμένοι είπαν ότι ο δικός χάρτης θα πρέπει να συνδεθεί περισσότερο με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ενδεχομένω ναι, αλλά ενδεχομένω να περιορίσει και αυτό τι φιλοδοξίε μα. Ενδεχομένω ορισμένα πράγματα να μην υπάρχουν στο δικό χάρτη και να θέλουμε παρόλα αυτά να τα επιτύχουμε στα πλαίσια του προγράμματο τη Στοκχόλμη. Ο δικό χάρτη αυτή τη στιγμή ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υπάρχει ένα πράσινο βιβλίο, μια πράσινη βίβλο για την κράτηση εγώ όμω θα ήθελα να έχουμε μία υπόσχεση, αν θέλετε, γι' αυτό, μία διασφάλιση ότι θα δούμε τελικά κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω πώς θα καταφέρετε με ξεχωριστές αποφάσεις πλαίσιο να, να περάσετε σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες στα όσα λέγονται στον οδικό χάρτη, αλλά είναι σημαντικό να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε όλες τις αποφάσεις πλαίσιο. και όντως αναγνωρίζω ότι πρέπει να γίνει από κάπου μια αρχή και είναι πολύ λυπηρό ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά τα οποία είναι υπαρκτά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό τελικά και για αυτό το λόγο να καταφέρουμε να έχουμε ένα συνολικό πρόγραμμα για την προάσπιση των δικαιωμάτων αυτό σε επαφές που είχαμε αρμοδίους στο Ηνωμένο Βασίλειο, άκουσα ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Πάρα πολλοί έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, ακριβώς επειδή δεν κατοχυρώνονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης όλα αυτά τα δικαιώματα του εναγωμένου. Και η κατάσταση σίγουρα θα επιδεινωθεί, Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Το Συμβούλιο έχει θέσει μια προθεσμία έχει ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλει την γνωμοδότησή του μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου και θα θέλαμε και το Συμβούλιο βέβαια να μας δώσει το έγγραφο το οποίο έλαβε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης και σας ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να αποχωρήσω και εγώ σε 10 λεπτά μου ζητήθηκε λίγο την τελευταία στιγμή να προεδρεύσω τη συνεδρίαση αυτή. Κάποιο άλλο λοιπόν θα πρέπει να με αντικαταστήσει. Α περάσουμε στο σημείο 29 τη ημερήσια διάταξη μεταφορά των διαδικασιών σε ποινικέ υποθέσει. Η κυρία Μπένοβα διορίστηκε σήμερα το πρωί συγγήτρια. Δυστυχώ απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Ο κύριο Μόερα όμω θα την αντικαταστήσει. Θέλετε να πάρετε τώρα το λόγο, να ακούσετε μάλλον πρώτα το Συμβούλιο. Να μα παρουσιάσει καλύτερα το Συμβούλιο πρώτα την κατάσταση. Κυρία Βέμπερ, εσείς θα πάρετε το λόγο. Σας ζητώ λοιπόν να είστε πραγματικά πάρα πάρα πολύ σύντομοι και δυνατόν να κάνετε μία σύνοψη των όσων θέλετε να μας πείτε γρήγορα αυτή τη στιγμή, περιληπτικά να μας τα πείτε, γιατί όλοι θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη, συνεργασία, τη σε αυτή εγκαίρωση και νωρίτερα. Πράγμα θα ήταν ιδιαίτερα επαναστατικό. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαστε δυνατόν πιο σύντομοι γίνεται. Σημείο φετηρία για την πρόταση αυτή για τη μεταφορά διαδικασιών σε ποινικέ υποθέσει είναι ότι δεν υπάρχει κοινό νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε μια σύμβαση του 1972 από το Συμβούλιο τη Ευρώπη, η οποία θα μπορούσε στην πράξη να λειτουργήσει, αλλά δεν υπάρχει καμία προβλεπόμενη κοινοτική διαδικασία για να γίνει αυτή η μεταφορά των διαδικασιών σε ποινικέ υποθέσει. Γι' αυτό το λόγο η Ειδική Προεδρία ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή, την οποία υποστηρίζουν 16 κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Στόχο εδώ πέρα είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα, ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη και το οποίο θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά μας κατά τη μεταφορά των διαδικασιών σε ποινικέ υποθέσεις διασφαλίζοντας επίσης τα δικαιώματα των ε, υπόπτων των ε, κατηγορουμένων. Προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα μεν, αλλά και ένα σύστημα το οποίο θα έχει συγκεκριμένε δικλείδε. αφού ήταν η Super Tour που η πιο γρήγορη παρουσίαση που μπορούσα να κάνω ποτέ. Σα ευχαριστώ πολύ και με σχέση σα για περισσότερε παρατηρήσει. Μα σα ευχαριστώ πολύ και γνωρίζω, είναι απόλυτα γνωστό ότι η Σουηδία είναι αποτελεσματική και σύντομη. Διερωτώ με, για ποιο λόγο φαίνεται τελικά ότι ε, οι εγκληματίες σε διεθνές επίπεδο είναι σε θέση να λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά και να συνεργάζονται τόσο καλά χωρίς να έχουν προβλήματα ούτε συνεννόηση ούτε επικοινωνία μεταξύ τους. κύριος Μωράης, δεν χρειάζονται ίσως διερμηνείς. Δεν το ξέρει κανείς αυτό τι γίνεται, αν δουλεύουμε διερμηνείς ή εγκληματίες. Ευχαριστώ, είναι πολύ σύντομη η παρουσίαση που ακούσαμε και εγώ θα είμαι σύντομος. Ζητώ συγγνώμη για το ότι η κυρία Μπένοβα απουσιάζει. Κάποια πολύ σύντομα στοιχεία τώρα, παρατηρήσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ως απόφαση πλαίσιο. Πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα όσον αφορά δικαιοδοσία στα κράτη-μέλη για να μην υπάρχει διπλή δίκη ενός ατόμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ε, ως θέμα και είναι λάθος το ότι υποχρεώθηκε να δουλέψει δύο φορές για δύο παρόμοια νομοθετήματα το Κοινοβούλιο. Είχαμε την έκθεση Βέμπερ σήμερα το πρωί και νέα πρόταση φαίνεται ότι έχει κάποιες επικαλύψεις όσον αφορά το εύρος. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, θα έπρεπε να εξηγήσουν περισσότερο πώς θα εξορθολογήσουν το νομικό πλαίσιο στην νομοθεσία σε σχέση με αυτά και με σκληρό τρόπο θα δουλέψει η κυρία Μπένοβα με τους κοιόδης εισηγητές για να επιληθούν αυτά τα θέματα. Ολοκλήρωσα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ένας συνάδελφος πίσω ζήτησε τον λόγο. Δεν μπορώ να διαβάσω το όνομά σας. Εσείς έχετε τον λόγο. Ήθελα να επισημάνω κάποιες παρατηρήσεις από πλευράς μου σε σχέση με αυτό το σχέδιο Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι ένα, πρόγραμμα, εγχείρημα πολύ ενδιαφέρον διότι πράγματι η αύξηση των διασυνοριακών εγκλημάτων και αδικημάτων σίγουρα θα μας υποχρεώσει να προβούμε σε μια ρύθμιση που θα επιτρέπει την αποφυγή του nec bis in idem, να μην υπάρχει διπλή δίκη για την ίδια υπόθεση. Χρειάζεται ένα μέσο το οποίο θα επιτρέπει η δίωξη, η ποινική δίωξη να γίνεται σε μία χώρα μόνο. Όταν αυτό το αδίκημα γίνεται πιο συχνά και μάλιστα επαναλαμβάνεται σε διαφορετικές χώρες. Τρεις παρατηρήσεις θα θέλα να διατυπώσω προ το Συμβούλιο, ευχαριστώντα για αυτό το σχέδιο από πλευρά του. Τρεις παρατηρήσεις που νομίζω είναι ενδιαφέρουσε. Η πρώτη παρατήρηση. Εγώ εκτιμώ πρέπει να πω θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη αμφισημία σε αυτό το εγχείρημα. Μεγάλη αμφισημία. Αληθεύει, δεν υπάρχει νομική βάση για το θέμα, αλλά υπάρχουν 16 χώρες που επιθυμούν να προχωρήσουμε. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, αυτό που θεωρώ είναι ότι είναι, αν θέλετε, μια διατύπωση, μια γλώσσα σε σχέση με την ε, σύμβαση, με τη ρύθμιση, που ε, δεν έχει εδώ κάποιο δεσμευτικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει ορολογία που να υποχρεώνει, ας το πω το κράτος που είναι είναι αποδέκτης ενός αιτήματο να δεχθεί το αίτημα αυτό. Εγώ από την άλλη πλευρά και με την απουσία συγκεκριμένης μορφής όσον αφορά διορίες και προθεσμίες. Στο άρθρο 13 για παράδειγμα, όταν η χώρα η οποία αποδέχεται να τεδέχεται ένα τέτοιο αίτημα πρέπει να απαντήσει σε άλλη χώρα που ζητεί, που θέτει αυτό το αίτημα και ζητεί να γίνει δίκη στη χώρα που αιτείται αυτό για ένα δίκημα που έγινε σε δύο ε, μέρη διαφορετικά πρέπει να απαντήσει. Ναι, πρέπει να απαντήσει αλλά δεν έχει προθεσμία η διορία. Πρέπει όμως άμεσα να απαντήσει και δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό να απαντήσει χωρίς καθυστέρηση. Τι ακριβώς συμβαίνει. Το ίδιο και στους λόγους που θεσπίζονται για τους οποίους μια χώρα μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια σε ένα αίτημα ώστε να είναι η άλλη χώρα εκείνη που θα αναλάβει την εκδίκαση μια υπόθεση. Μπορεί να υπάρχει ένας μεγάλος μεγάλο αριθμό λόγων για να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Όμω, με ανησυχεί ότι στην πρακτική εφαρμογή αυτό το σύστημα δεν χρησιμοποιείται θετικά διότι δεν απαντούν θετικά στα αιτήματα αυτά οι χώρε που δέχονται τέτοια αιτήματα. Με την άποψη τη εθνική επικυριαρχίας, δηλαδή είναι δική μου αρμοδιότητα αυτή και όχι δική σου στην δικαιοδοσία. Και έτσι δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Γι' αυτό δεύτερο στοιχείο, για να προχωρήσουμε στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων όταν έχει, υπάρχει άρνηση της χώρας από να δεχθεί το αίτημα άλλης χώρας για την διεκδίκαση ε, μιας υπόθεσης ε, στη χώρα αυτή, τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση. Κανείς δεν επιλύει τέτοια θέματα. Με ανησυχεί εν τέλει στο άρθρο 4 για την αναφορά σε μη δικαστικές αρχές που απαιτεί συγκεκριμενοποίηση, εξειδίκευση. Γιατί όταν κάνουμε λόγο για αρχές που δεν είναι ομοιογενείς εδώ, όταν για μια χώρα που δίνει συνέχεια σε τέτοιου είδους θέματα δεν είναι οι δικαστικές αρχές, ποιε είναι άλλοι δικαστές άλλη άλλης ε, δεν θα ε, εμπιστευτούν να επομιστούν αυτή την υπόθεση. Είναι θέματα που πρέπει να επιληθούν, να εξειδικευτούν στην έναρξη αυτής της συζήτησης. Φυσικά μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο αυτά τα πράγματα στο μέλλον με τροπολογίες ή βελτιώνοντας αυτό το κείμενο το οποίο το εκτιμώ θετικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλετε να παρέμβετε σύντομα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα μιλήσω εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για πρωτοβουλία των κρατών μελών, όπως ξέρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή. Θεωρούμε και εμείς ότι αποσιάζει τέτοια νομοθεσία στο ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά τις συνεργασίες, ποινικέ διαδικασίες μεταξύ των κρατών μελών. Είμαστε λοιπόν υπέρ της πρότασης αυτής, αρκεί βέβαια να επιφέρει μια προστιθέμενη αξία. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής η υφιστάμενη πρόταση αποτελεί προστιθέμενη αξία γιατί δημιουργεί κοινού κανόνες που θα ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη. Μέχρι στιγμής μόνο 13 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επικυρώσει και εφαρμόζουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι όντως χρειαζόμαστε ένα νέο νομικό μέσο το οποίο ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα τα ερωτήματά σα, θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ αρχής είχε πει ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένους κανόνες και χρειαζόμαστε και προθεσμίες. Είπαμε πολλές φορές και σε συνεργασία με πολλά άλλα κράτη-μέλη όπως με το Βέλγιο ότι πρέπει να αλλάξει η διατύπωση του άρθρου 13, η οποία τροποποιήθηκε. Η νέα διατύπωση δεν προβλέπει προθεσμία, αλλά λέει ότι οι αρμόδιες αρχές εθνικές θα θέσουν τις προθεσμίες αυτές. Μόνο και μόνο αυτό από μόνο το αποτελεί πρόοδο. Και εντοπίζεται βέβαια και οποιαδήποτε καθυστέρηση ως πρόβλημα στην συνεργασία που θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε λοιπόν εμείς να εξασφαλίσουμε σε κάθε περίπτωση ότι η πρόταση αυτή θα επιφέρει προς τη θέμενη αξία. Μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται επιτυχάνεται αυτό από την πρόταση. Ελπίζω απλώς ότι στο βωμό της ομιμορφίας δεν θα θυσιαστεί αυτή προς τη θέμενη αξία που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Προθεσμία που έχει θέσει το Συμβούλιο για την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η 17η Δεκεμβρίου και σας πενθυμίζω ότι η συγγήτριά μας είναι η κυρία Μπένοβα. επειδή αντικαθιστώ τον πρόεδρο και εγώ ίδια πρέπει να αποχωρήσω, θα μπορούσα να ζητήσω από το πρεσβύτερο μέλος της Επιτροπής μας, που είναι ο κύριος Διόγκ, αν θα είχε την... αν μου την τιμή να έρθει να με αντικαταστήσει. Ευχαριστώ. Uh, λοιπόν, με εκπλήσει το να βρίσκομαι εδώ ως πρόεδρος, εντάξει, αλλά... Λοιπόν, σημείο 31. Η δημιουργία ενός δικτύου πρόληψης εγκλήματος. Πρώτα μια σύντομη παρουσίαση από τη Σουηδική Προεδρία, λοιπόν, επ' αυτού. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο εισηγητής. Λοιπόν, η Σουηδική Προεδρία πρώτα. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πάλι εγώ, λοιπόν κάνοντας λόγο γι' αυτό, θα πρέπει να είμαι σύντομη υποθέτω. Λοιπόν, ίσως εδώ όχι τόσο σύντομη όσο και προηγούμενα, αλλά παρόλα αυτά, για να σκιαγραφίσω και να πω ήταν μια πρωτοβουλία που ανελήφθη από ένα αριθμό κρατών μελών. Εδώ 11 κράτη-μέλη ανέλαβαν την πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία αυτή έγινε, ανελήφθη με βάση <clears throat> μια αξιολόγηση, μια αποτίμηση που έγινε με βάση το σημερινό δίκτυο πρόληψης εγκλήματος που ταυτοποίησε και εντόπισε έναν αριθμό ελλείψεων και αδυναμιών για το πώς λειτουργεί το δίκτυο αυτό σήμερα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε, αποκινούμε έναν αριθμό άλλων κρατών μελών, αναλάβουμε πρωτοβουλία να κάνουμε μια επιδιόρθωση, επανόρθωση του συστήματος, να διορθώσουμε τις αδυναμίες για να ενδυναμώσουμε το, την UCP ε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Το UCPN ε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος και να ξεκινήσουμε επικεντρωνόμενοι σε τρεις άξονες, σε τρία θέματα. Πρώτον, να τονίσουμε περισσότερο τον ρόλο των κρατών μελών μέσα στο ίδιο το δίκτυο. Είναι ένα δίκτυο για τα κράτη-μέλη λοιπόν αυτό. Και είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη και οι συνεισφορές τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο δίκτυο το ίδιο μπορούν να ενισχυθούν, να ενδυναμωθούν. Πρώτη παρατήρηση αυτή για την πρόταση. Δεύτερη παρατήρηση. Η πρόταση είναι να επικεντρώσουμε τη δουλειά στο EUCPN, στο Ευρωπαϊκό, όπω είπα, Δίκτυο Πρόληψη του Εγκλήματο και να υπάρξει πρόσθετη αξία, όφελο που θα δημιουργηθεί στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε λοιπόν, να το πω έτσι, μια σύμπτυξη, μια πιο αποτελεσματική διάρθρωση των θεμάτων στα οποία θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε. Τρίτο σημείο, εξίσου σημαντικό, να προσπαθήσουμε και να βρούμε μια λύση για τη γραμματεία, το ζήτημα της γραμματείας που εντοπίστηκε, ταυτοποιήθηκε από αυτή την αποτίμηση ως μια δυναμία στο σύστημα. Δεν, υπάρχει ε, γραμματεία. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία και οι κύριες ιδέες πίσω από αυτήν την πρόταση που αυτή τη στιγμή συζητείται και εξετάζεται από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τις δομές αυτές. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια εξίσου σύντομη παρουσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε πέρυσι μια πλήρη αξιολόγηση και αναθεώρηση του δικτύου αυτού, όπως είπε και εκπρόσωπος ειδική Προεδρίας. Κάναμε μια πολύ πλήρη έκθεση, έχουμε μια πολύ πλήρη έκθεση με συγκεκριμένε συστάσει και χαιρόμαστε πολύ που πολλέ από τι συστάσει αυτέ αντικατοπτρίζονται τώρα στο κείμενο τη Προεδρία και των κρατών μελών. Πρέπει να σα πω όμω ότι η τελική τοποθέτηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Αυτό θα πρέπει να γίνει από το Κολέγιο των Επιτρόπων και θα γίνει συγκεκριμένα τον Οκτώβριο κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ήδη μπορώ να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα υπέρ της χρηματοδότησης του δικτύου αυτού μέσω σύμβασης δημόσιας παροχής και πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε δεσμεύσει 900.000 ευρώ, πολύ σημαντική αύξηση σχέση με τα ποσά που είχαμε δεσμεύσει στο παρελθόν για το δίκτυο αυτό. Τούτο λεχθέντον τώρα, θα πρέπει να υπάρχει μια συνένεση των κρατών μελών για το εφιστάμενο κείμενο, το οποίο αναφέρεται σε πάλι συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα πρέπει να δοθεί στο δίκτυο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, κάνει, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να είναι δυνατόν να δοθεί χρηματοδότηση στο δίκτυο αυτό μέσω ενός ποσού που θα δοθεί για τη χρηματοδότηση του δικτύου αυτού. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής από δημοσιονομικής ή νομικής πλευράς δεν έχουμε εντοπίσει κανένα πρόβλημα με το κείμενο το οποίο τυχαίνει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ και για την συντομία και τη σαφηνία σας. Τώρα θα λάβει τον λόγο ο εισηγητής που είναι η κυρία Σόνια Αρφάνο, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Σουηδική Προεδρία και την Κομισιόν. Εγώ άκουσα όλες τις παρουσιάσεις. Η Προεδρία είπε ότι θα πρέπει να δώσουμε μια μεγαλύτε, ένα μεγαλύτερο ρόλο και δημοσιότητα στα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν είπε ότι δεν υπάρχουν οικονομικά και νομικά προβλήματα. Εγώ όμως δεν άκουσα να γίνεται αναφορά στο πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι αν αυτή είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στην εγκληματικότητα, είναι μία απάντηση εντελώς ανεπαρκής. Δηλαδή φαίνεται ότι τελικά έχουμε εδώ μία διάρθρωση που την έχουμε εκεί γιατί έχουμε λεφτά και θέλουμε να τα ξοδέψουμε. Δεν δούλεψε ποτέ αποτελεσματικά. Υπάρχει μία γραμματεία, ένας υπάλληλος και μία ερευνήτρια part-time. Για να μπορέσουμε να έχουμε παρακολούθηση και καταγραφή των εγκλημάτων ε, αυτό είναι εντελώς ανεπαρκές. Υπήρχε και ένα φόρουμ το οποίο δεν έκανε τίποτα. Και έχω επίσης και μια άλλη εντύπωση, ακόμη χειρότερη από την προηγούμενη, ότι δηλαδή η καταπολέμηση του εγκλήματος θεωρείται σε δεύτερη κατηγορία από ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εγώ δεν θέλω να κάνω εδώ μία ταξινόμηση ε, του πόσο σοβαρή είναι η τρομοκρατία, πιο σοβαρή η τρομοκρατία ή η εγκληματικότητα. Εμείς διαπιστώνουμε καθημερινά ότι η εγκληματικότητα έχει παρισφρήσει απόλυτα σε κρατικά συστήματα. Πράγμα που η τρομοκρατία δεν είμαστε σίγουροι ότι το έχει κάνει. Όταν εμείς μιλάμε για τρομοκρατία δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι υπάρχει σωματεμπορία. Αλλά η διακίνηση των ναρκωτικών, το ξέπλυμα του βρώμικου κρίματος, τα διαχειρίζονται το οργανωμένο ε, έγκλημα. στα ναρκωτικά και στο ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος η απάντηση που δίνει η Ευρώπη είναι αυτή, ε, πραγματικά μου φαίνεται εντελώς ανεπαρκής. Τι έκανε το δίκτυο για να... για την πρόληψη του εγκλήματος. Το δίκτυο επίσης αμφισβητήθηκε πάρα πολλές φορές. Πώς θα το λύσουν λοιπόν το Συμβούλιο και η Κομισιόν το θέμα. Από ό,τι άκουσα το Συμβούλιο θέλει να τα δώσει όλα αυτά ε, σε έναν εξωτερικό οργανισμό να τα διαχειριστεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πει να διευρύνουμε τον ορισμό ε, για, του οργανωμένου εγκλήματος όλα αυτά γιατί αγνοήθηκαν. Και γιατί η δραστηριότητα του δικτύου είναι μυστική. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Διότι αν αυτή τελικά είναι η πραγματική ευκαιρία να αναδιαρθώσουμε το δίκτυο, να δώσουμε μία υπόσταση σε αυτόν τον οργανισμό, ε, είναι ευπρόσδεκτη. Κυρία Μακαβόη. Ευχαριστώ. Είμαι σκιώδη συγγήτρια για το ΕΛΚΑ. Χαίρομαι πολύ που είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Αλφάνο. Από ό,τι κατάλαβα, η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την πρόληψη του εγκλήματος, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι το έγκλημα αυτό θα μπορούσε να προκύψει κάπου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ προσπαθώ μέσω του δικτύου αυτού να το σταματήσω. Θα ήθελα να γνωρίζω εγώ ποια είναι προστιθέμενη αξία, απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για ποιο λόγο θα λειτουργήσει αυτή τη φορά το δίκτυο τη στιγμή που δεν έγινε κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Βέμπερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από το τέλος, προσπαθώντας να απαντήσω στον τελευταίο ερώτηση. Για ποιο λόγο θα επιτύχουμε αυτή τη φορά. Κοιτάξτε, όλη αυτή η διαδικασία, το ότι κάνουμε δηλαδή μια συζήτηση για το EUCPN, ότι προσπαθούμε να δούμε ποια θα είναι η προσθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος, για ποιο λόγο πρέπει να έχουμε διαδίκτυο κτλ. Όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ θετική γιατί ε, ουσιαστικά κάνει και τα ίδια τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν περισσότερο και να ξεκινήσουν και αυτά μια συζήτηση για το πώς θα πρέπει να διαρθρωθεί το δίκτυο και πώς θα πρέπει να λειτουργήσει. Απομένει να δούμε βέβαια θα λειτουργήσει αυτή τη φορά αλλά σίγουρα το όλο εγχείρημα μέχρι στιγμή ήταν πολύ θετικό, γιατί αν μη τι άλλο εμπλέξαμε συζήτηση περισσότερο τα κράτη-μέλη, τα οποία τώρα ενδιαφέρονται και λένε και τη γνώμη του πώ θα πρέπει να λειτουργεί αυτό το δίκτυο. Είναι πολύ θετική η ανταπόκριση, αν μη τι άλλο, που είχαμε στη συζήτηση αυτή για το δίκτυο αυτό. Τώρα, όσον αφορά την μυστικότητα στην οποία αναφερθήκατε στα πλαίσια της λειτουργίας του δικτύου, δεν κατάλαβα πολύ καλά το ερώτημά σας. Δεν πρόκειται για ένα μυστικό δίκτυο. Είναι ένα δίκτυο το οποίο απαρτίζεται από μέλη που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη και προφανώς στα πλαίσια του δικτύου αυτού προβλέπεται επικοινωνία με τους ε, εκπροσώπους του. Θα υπάρχει μάλιστα μια ιστοσελίδα που θα παρουσιάζει τις εργασίες του δικτύου. Δεν τίθεται ζήτημα δηλαδή μυστικότητας. Σαφώς θα μπορούσε να βελτιωθεί βέβαια το εφιστάμενο σύστημα ενημέρωσης που έχει το δίκτυο, προκειμένου να ενημερώνεται καλύτερα ο κόσμος για τις εργασίες του. Και πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο, εφόσον γίνει αναθεώρηση αυτή, θα έχει και το δίκτυο ένα μεγαλύτερο επίπεδο διαφάνειας. Ελπίζω να απάντησα έτσι στην ερώτησή σας. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα επικεντρωθώ στι ερωτήσει από πλευρά εισήγηση όσον αφορά την χρηματοδότηση. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή δώσαμε κατά τα τελευταία δύο έτη 180.000 ευρώ για την λειτουργία του δικτύου και πιο εξειδικευμένα στην οργάνωση για τις, ε, την διάσκεψη για τις βέλτιστες πρακτικές ε, και για το έπαθλο πρόληψης ε, εγκλήματος, εγκληματικότητας. Για να δώσουμε μεγαλύτερο, περισσότερο ευδιάκριτο χαρακτήρα σε αυτό το δίκτυο. Όσον αφορά τα όσα γίνονται δημοσιονομικά για το 2010, εγγράψαμε στο πρόγραμμα εργασίας μας 900.000 ευρώ. Πρέπει να τονίσω ότι το ετήσιο πρόγραμμα πρέπει ακόμα να εγκριθεί είναι η στοχοθέτηση, η ημερομηνία για έγκριση 9 Οκτωβρίου. Όπω είπα, ενεγράφει αυτό υπό τον τίτλο Δημοσίων Προμηθειών. Και δεν θέλω να επισέλθω τώρα σε τεχνικά θέματα και νομικές λεπτομέρειες Ίσως όμως η πιο σημαντική επίπτωση αυτού του τρόπου χρηματοδότησης του δικτύου θα είναι ότι θα έπρεπε να είναι ότι οι δραστηριότητες θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα απαιτείται από τα κράτη-μέλη κάποια ε, συνεισφορά και έτσι λοιπόν θα πρέπει αν όταν και όταν αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Σαβόνας θα παρέμενε επίσημα επικεφαλής της Γραμματείας ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε όμως να κάνουμε outsourcing, να δοθεί προς τα έξω η εντολή ανάληψης αυτών των αρμοδιοτήτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν μερικής απασχόλησης, ένα μερικής απασχόλησης άτομο που καλύπτει τις ανάγκες. Θα μπορούσε να αυξηθεί το προσωπικό σε τρία ή τέσσερα μέλη για το δίκτυο αυτό. Το σημερινό ενισχύει κείμενο προβλέπει μια χορήγηση ε, κεφαλαίου για την λειτουργία. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βρουν μια δυνατότητα συγχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του δικτύου. Γιατί μια χορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί ποτέ να καλύπτει 100% του κόστους. Δεν θα υπάρχει διοικητική διασύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραμματείας ε, του δικτύου και σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, τη συμμετοχή σε εξωτερικά όργανα θα συμμετέχει στο έργο του, δικτύου αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρατηρητής. Πράγμα που θα σημαίνει ότι δεν θα είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχει σε συζητήσεις για το διοργανωτικό, τη διοργανωτική διάρθρωση ή τη χρηματοδότηση του δικτύου για να αποφευθεί σύγκρουση δραστηριοτήτων. Θα είναι σε θέση όμως επί της ουσίας να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις απόψεις για τις πολιτικές πρόληψεις του εγκλήματος. Ευχαριστώ. Δεν γνωρίζω αν θα ήθελε να επανέλθει και να παρέμβει η συγγήτρια μετά από τις παρεμβάσεις του Συμβουλίου και της, Ευρωπαϊκή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είμαι πολύ σύντομη. Εγώ περίμενα πιο σαφείς ερωτήσεις. Το θέμα για μένα δεν είναι ε, η δημοσιότητα, η ορατότητα του δικτύου Εγώ πιστεύω απλώς ότι είναι απαράδεκτο μόνο δύο-τρεις άνθρωποι να ασχολούνται με την περιφρούρηση και την παρακολούθηση του εγκλήματος. Θα έπρεπε να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να κάνουν την παρακολούθηση αυτή. Είναι εντελώς ανεπαρκές αυτό το σύστημα για την παρακολούθηση. Δεν πρόκειται ποτέ να περιφρουρήσουμε εμεί το έγκλημα κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εμείς παρακολουθούμε το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο φύγει άμεσα και τις 27 χώρες. Και απαιτούμε αυτή τη δουλειά να την κάνει μία γραμματεία με 1,5 άτομο προσωπικό. Είπαμε, δεν είναι ένα θέμα ορατότητας, είναι απλώς το πώς θα πρέπει να αλλάξουμε αυτό το δίκτυο αν θέλουμε πραγματικά να γίνει λειτουργικό. Σίγουρα υπάρχει το δίκτυο, υπάρχει η ιστοσελίδα την είδα, αλλά δεν καταλαβαίνω σε τι μπορεί να βοηθάει και δεν έδωσε και ποτέ λογαριασμό κανείς για τίποτα στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω με οι συζητήσεις που θα γίνουν μεταξύ συγγήτριας και σκιωδών συγγητών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πεπισμένο για την αποτελεσματικότητα της πρότασης αυτής και προφανώς θα υπάρχουν περισσότερες συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλει κανεί άλλο το λόγο, να σα πω ποιε είναι οι προθεσμίε. Δεν υπάρχει ακόμα προθεσμία. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Το επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης ε, για τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα έχει αναβληθεί. Περνάμε στα διάφορα. Δεν νομίζω ότι έχουμε τίποτα στα διάφορα, έτσι δεν είναι. Καμία ανακοίνωση, επομένω λύεται τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ.